Colleghi, buongiorno. Καλημέρα σα Να ξεκινήσουμε με την ε, τελευταία τμήμα τη συνεδρίασή μα. Χθε ήταν ε, εντατική η ημέρα και ολοκληρώσαμε με την ακρόση του κυρίου Τσότη, ο οποίος ε, μας έδωσε την αίσθηση ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών ε, για την υποστήριξη των θυμάτων ε, και για την καταπολέμηση της μαφίας όπως ε, και ο ίδιος ο ρόλος κοινωνίας των πολιτών ενισχύεται από αυτή την καταπολέμηση της μαφίας σήμερα. Συνεχίζουμε αυτή τη διαδρομή γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι δεν είναι δυνατόν να θέσουμε την τον αγώνα για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματο μόνο στι διοικητικέ και στι δικαστικέ αρχέ, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών ε, είναι ζωτική σημασία. Είναι ρόλο κλειδί. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μπέρνφινκερ, ο οποίο είναι επικεφαλή τη αστυνομία του Βερολίνου, ο οποίο ε, συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματο και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φόρτε που εκπροσωπεί το δίκτυο Φλερ. Έχουμε δύο πραγματικότητες, ε, μία θεσμική πραγματικότητα, ε, ενώ έχουμε και έναν εκπρόσωπο που θα μας εξηγήσει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, όμως κατανοούμε πως αυτές οι δύο πραγματικότητες ε, μπορούν να συμβαδίζουν. Η συζήτηση θα ακολουθήσει ό,τι κάναμε και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή δύο μιλητές θα έχουν 15 λεπτά για την παρουσίασή τους, κατόπιν θα πάρουν το λόγο ο συγητής, οι συντονιστές και οι συνάδελφοι για δύο λεπτά και κατόπιν θα ξαναδώσουμε το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν στα σχόλιά σας και στις ερωτήσεις σας. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως και θα δώσω το λόγο στον κύριο Φίνγκερ. Παρακαλώ. Um, uh, Καλημέρα σας. Είμαι ο Πέρντ Φίγκερ και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εδώ και 43 χρόνια ε, είμαι αστυνομικός. Το θέμα με το οποίο ασχολούμαι είναι το οργανωμένο έγκλημα, ε, τα εγκλήματα που διαπράττουν οι συμμορίες. Εγώ λοιπόν είμαι αρμόδιος για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο Βερολίνο. Η δική μου υπηρεσία είναι στη Γερμανία η κύρια ε, υπηρεσία η οποία διεξάγει τον αγώνα της ε, αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να μιλήσω γερμανικά, αν δεν έχετε αντίρρηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. κατά την επέτειο της 20ης επαιτίου της δολοφονίας του Τζοβάνι Φαλκόνε και του Πάολο Μπορσελίνο ξεκινάω με ε, μια εισαγωγή για να σας παρουσιάσω τη θέση της υπηρεσίας μου, τη θέση τη δική μας της αστυνομίας του Βερολίνου ε, για αυτά τα θέματα. Για μας ε, η αντιμετώπιση του εγκλήματος σημαίνει προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κράτος έχει το καθήκον να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Το κράτος λοιπόν πρέπει να αναλαμβάνει δράση οποτεδήποτε απειλούνται αυτά τα δικαιώματα το, ο άνθρωπος, ε, όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μην υφίστανται καταπίεση, εκμετάλλευση, να έχουν πρόσβαση σε κατοικία και σε άλλες βασικές ε, ανάγκες, κάλυψη βασικών αναγκών. Θα ήθελα λοιπόν συνεχίζοντας να σας πω το εξής το έγκλημα και κυρίως το οργανωμένο έγκλημα έχει λάβει μια οργανωμένη, παγκοσμιοποιημένη μορφή και ε, απειλεί τους ανθρώπους, ε, καταστρέφει τις ε, θέσεις εργασίας τους ε, κατοίκους, τους πολίτες, ε, τους ε, εκφοβίζει, παρεμποδίζει την ελευθερία έκφρασης γνώμης, παρεμποδίζει την διαφάνεια και αφήνει τους ανθρώπους την τύχη τους, ενώ παράλληλα παρατηρείται ότι μεγιστοποιείται ο προσπορισμός κέρδους από πλευράς συμμοριών. Δυστυχώς με τον τρόπο αυτό καταστρέφεται η δυνατότητα ίσων ευκαιριών παρατηρείται απληστία, καταστρέφεται το περιβάλλον και η ελευθερία έκφρασης γνώμης, η ελευθεροτυπία και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους αμέτρητους φόνους δημοσιογράφων και πολλών άλλων ανά τον κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει μόνο στις ε, φτωχές χώρες, σε χώρες όπου δεν υφίσταται δημοκρατική παράδοση. Το φαινόμενο αυτό είναι βαθιά ριζωμένο και μέσα στην ίδια την καρδιά της Ευρώπης, ακόμα και στη Γερμανία, όπου στη Γερμανία ειδικά τα μέλη της ε, μαφίας επικαλούμενοι το Σύνταγμα ε, δικάζουν και καταφέρουν στα δικαστήρια για να καταδικάσουν, εφόσον το επιτύχουν, ε, όσους είναι εκφραστές της ελευθεροτυπίας. Αν όμως δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών, δεν υπάρχει και νομιμοποίηση του κράτους και δεν υπάρχει η διάδοση του πολιτισμού της νομιμότητας. Το κράτος ε, δικαίου εκφράζεται μέσα από το κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου και κοινωνικό κράτος αλληλοσυμπληρώνονται. Ο δικός μας λοιπόν αγώνας για τη νομιμότητα είναι δυνατόν να κερδιθεί μόνο εφόσον συνδυαστεί με τον αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη και επίσης ε, και με την προστασία ε, του περιβάλλοντος από λαιλασίες και καταστροφές. Άρα δηλαδή πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε βοηθήσουμε τους αδύναμους, να τους δώσουμε φωνή, να εισακουστεί η φωνή τους, γιατί πολλές φορές κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ε, προς όφελος οικονομικών ε, συμφερόντων η Occupy the Wall Street Bebegung, ε, υπάρχει αυτή η κίνηση όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εκεί λοιπόν οι περισσότεροι λένε ότι επιθυμούν να συνενώσουν τις ε, δυνάμεις τους, ε, επιθυμούν να υπάρχει πολυφωνία και αυτό ως ευκαιρία ενός δημοκρατικού πλουραλισμού. Επίσης πολλοί επιθυμούν να υπάρχει αλληλεγγύη αλληλεγγύη κατά όλων των ε, μορφών εκμετάλλευσης ε, ανθρώπου από άνθρωπο. Κάτι τέτοιο αφορά κυρίως το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα είναι εκείνο ε, το οποίο διαδίδει τέτοιου είδου πρακτικέ. Μόνο από κοινού το κράτο και η κοινωνία των πολιτών έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα ως αστυνομικός ε, ε, ε, μιας πρωτεύουσας της Ευρώπης, του Βερολίνου, μιας πρωτεύουσα κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναφέρω και κάποια πρακτικά στοιχεία. Ακούσαμε πάρα πολλά για συγκλονιστικά στοιχεία για συγκλονιστικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσει το οργανωμένο έγκλημα. Και τώρα θα ήθελα εγώ να σας παρουσιάσω κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό, που δείχνει ότι από κοινού μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει διέξοδος εφόσον ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Και θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω την κατάσταση στο Βερολίνο και ποιες ακριβώς είναι οι εξελίξεις. Σε αντίθεση λοιπόν με ε, πάρα πολλές ε, δημοσιεύσεις ε, στον τύπο που αφορούν ε, στην Ιταλική μαφία ότι δήθεν η Γερμανία έχει παραμελήσει το θέμα αυτό. Ήδη κατά τη δεκαετία του 80 ε, συστήθηκε ε, μια ανακριτική ομάδα στο Βερολίνο η οποία επιλήφθηκε ιδιαίτερα ακριβώς αυτής της μαφίας της Ιταλίας. Στις αρχές του 2000 συστήσαμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για οργανωμένο έγκλημα στο Βερολίνο λοιπόν και γενικότερα στη Γερμανία εκπονήσαμε μία μελέτη αξιολόγησης η οποία ασχολείται με την οργανωμένη εγκληματικότητα κυρίως με τη μορφή μαφίας. Ε, γνωρίζετε πολύ καλά την 15η Οκτωβρίου 2007 όπου είχαμε επτά δολοφονίες στο Duisburg της Γερμανίας. Αυτά που αναφέρθηκαν ε, την επόμενη μέρα ε, στον τύπο μπορείτε όλοι σας ε, να τα διαβάσετε. Οι οικογένειες των θυμάτων στη Γερμανία ανέφεραν ότι έχουν υποψίες για οργανωμένο έγκλημα στη Σουτγάρδη, σε άλλες πόλεις και στο Βερολίνο. Εμείς λοιπόν ε, τα δικά μας τα συμπεράσματα του Βερολίνου τα συγκρίναμε και με ε, ε, ερευνητικά συμπεράσματα άλλων πόλεων και πράγματι διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν μαφιόζικες οργανώσεις, η Καμόρα, η Ντραγκέτα, η Κοζανόστρα, οι ομάδες αυτές ασχολούνταν την εποχή εκείνη κυρίως ε, με ε, κλεμμένα αυτοκίνητα και με παραχαραγμένα νομίσματα, ε, χρηματονομι... παραχαραγμένο χρήμα κυρίως. Δεν υπήρχαν όμως συγκεκριμένα στοιχεία για τα θύματα του Βερολίνου. Την ίδια λοιπόν ημέρα διαβάσαμε στον τύπο στη Γερμανία ότι η Δραγκέτα κυρίως, είχε στο Βερολίνο 30 εστίες, οι οποίες εστίες όμως ήταν ε, λάθος, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, διαψεύστηκε αυτό και στον τύπο. Επειδή όμως καταρχήν έγινε λόγος για 30 εστίες της Δραγκέτα στο Βερολίνο, στην αρχική φάση, στο Ντούισμπουργκ, οι άνθρωποι αισθάνθηκαν όπως ακριβώς και στο Βερολίνο. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς ε, στο Βερολίνο είμαστε η πρωτεύουσα της πολιτικής, άρα δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει μας στείγει άμεσα. Κατόπιν, μετά από μεταγενέστερη αξιολόγηση και άλλων διεθνών στοιχείων, καταλήξαμε στο ότι ειδικά για το Βερολίνο δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο μετά από αυτές τις δολοφονίες που διαπράχτησαν στο Ντουισμπορκ θεωρήσαμε ότι όπως σας είπα εμείς δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο ε, να αντιμετωπίσουμε στο Βερολίνο. Αποφασίσαμε όμως παρόλα αυτά στις 28 να οργανώσουμε μια συνέντευξη τύπου γιατί ε, διαβάσαμε στις γερμανικές εφημερίες ότι οποιοδήποτε πάει στην πιτσερία και αγοράζει μια πίτσα αυτομάτως ε, συνεισφέρει ε, για την μαφία και ξαφνικά στη Γερμανία αισθάνθηκαν όλοι οι Γερμανοί ότι όλοι οι Ιταλοί είναι Αυτό όμως δεν μπορούσαμε να το επιτρέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ως ε, επικεφαλής ε, της αστρομικής διεύθυνσης του Βερολίνου βγήκα στα μέσα ενημέρωσης και είπα ότι αυτή την γενικευμένη υποψία απέναντι στους Ιταλούς τη διαψεύδω. Εγώ προστατεύω την Ιταλική κοινότητα από τέτοιου είδους κατηγορίες. Ε, θέλω να υπάρχει διαφάνεια, ε, όμως χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς να υποτιμούμε την εγκληματικότητα της μαφίας. Πράγματι, είπα, στη Γερμανία υπάρχουν ε, διαδικασίες αλλά και ε, διάφορες διασυνδέσεις της Δραγκέτα, της Καμόρα, της Κοζανόστρα. Και είπα επίσης ότι η γερμανική αστυνομία θεωρεί ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να υπάρχει να υπάρχουν ενημερωμένοι πολίτες, ενημερωμένοι επιχειρηματίες που συνεργάζονται με την αστυνομία. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο οχυρό ή οχύρωση απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, λίγες μέρες αν θέλετε μετά το Duisburg, ε, καταρτήσαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο προληπτικό γιατί ε, είπαμε τότε ότι το να έχουμε ένα σχέδιο στεγάνωσης αυτό δεν σημαίνει ομερτά για την ε, αστυνομία. Θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει, να μας δίνει πληροφορίες για να αντιμετωπίσουμε όλοι το οργανωμένο έγκλημα. Την επόμενη ημέρα χωρίς την δική μας παρέμβαση στο Βερολίνο με μια ε, συνέντευξη ε, τύπου ε, προέκυψε μια πρωτοβουλία που έλεγε «Μαφία, όχι σας ευχαριστώ». Μια Ιταλίδα προείστατο αυτής της πρωτοβουλίας και ακολούθησαν έξι Ιταλοί εστιατόρες, οι οποίοι με, με το μοντέλο που είχαμε χρησιμοποιήσει και εμείς ε, για την πίτσα είπαν ότι αυτοί δεν καταβάλουν προστασία στη μαφία. Είπαν ότι ως Ιταλοί ε, νιώθουν συγκλονισμένοι από τις δολοφονίες ε, στο Ντουισμπουργκ και είπαν επίσης ότι δηλώνουν ότι αποστασιοποιούνται από τέτοιου είδους ενέργειες. Το δήλωσαν μάλιστα κατηγορηματικά. Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς τέτοιου είδους συνεργασία έψαχνα να βρω. Στις 29 8 λοιπόν καταλήξαμε σε μια συμφωνία μια συμφωνία. Εγώ βεβαίως εκπροσωπούσα την δική μου την αρχή, την αστυνομική διεύθυνση. Εγώ ήμουν ο εκπρόσωπος ε, της ε, επιβολής του νόμου και ε, αυτή η δήλωση που βλέπετε, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε, είναι σύντομη, αλλά σας είπα, από τη μια πλευρά ήμουν εγώ και από την άλλη η επικεφαλής πρωτοβουλίας, η κυρία Γκραβίνη ε, νομίζω λεγόταν. Αυτά στις 29 Αυγούστου, 14 ημέρες μετά τις δολοφονίες στο Ντουισμπουργκ, είχαμε κατορθώσει στο Βερολίνο να συμμαχίσουμε και να αναλάβουμε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία με την Ιταλική κοινότητα. Μετά λοιπόν ε, βγήκαμε επιθετικά στον τύπο, είπα είπαμε, δείχνουμε όλοι το πρόσωπό μας στη μαφία. Η αστυνομία ε, μάλιστα προέβλεψε και για μια κόκκινη γραμμή, έναν τριψήφιο αριθμό. Ε, αυτό τον αριθμό τον γνωστοποιήσαμε σε όλους. Επίσης ε, ευαισθητοποιήσαμε το 100 όπως λέμε, τις αστυνομικές περιπόλους ε, μοιράσαμε διάφορα ενημερωτικά δελτία, χρησιμοποίησαμε το διαδίκτυο. Ε, στην ε, πόλη εμφανίστηκαν πάρα πολλά αυτοκόλλητα με αυτή την πρωτοβουλία της πίτσας και σήμερα υπάρχουν αυτά και είχαμε και πάρα πολλές από κοινού συζητήσεις. Όσοι λοιπόν ήθελαν να έρθουν σε επαφή με αυτή την ε, πρωτοβουλία έπρεπε να έρθουν σε επαφή με την κυρία Γκαβίνη μετά ε, μέσω αυτής με μένα και έτσι λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα μέσα από αυτή την πρωτοβουλία να έρθει κανείς άμεσα σε επαφή με την αστυνομία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί γνωρίζουμε πάρα πολλούς ε, όχι μόνο Ιταλούς αλλά και άλλους πολίτες από άλλες χώρες οι οποίες έχουν δυσκολία να έρθουν σε επαφή με τις αστυνομικές αρχές και να απευθυνθούν ε, και στην γερμανική αστυνομία. Μετά από έξι περίπου μήνες ε, είχαμε και την, ε, το πρώτο τεστ, την πρώτη δοκιμασία. Εμφανίστηκαν επτά απειλητικές επιστολές κατά 7 εστιατορίων. Ε, στο Βερολίνο, μην ξεχνάτε, έχουμε 3,5 εκατομμύρια κατοίκους ε, και έχουμε και πολλούς άλλους που δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένοι, δηλαδή μιλάμε για 4 με 5 εκατομμύρια κατ' ουσίαν. Στον τομέα αυτό εμφανίστηκε η απειλητική επιστολή κατά των Ιταλών επιχειρηματιών κατεβλήτησαν προσπάθειες ε, για να πάρουν προστασία, έγιναν πολλοί εμπρισμοί και οι ε, δράστες ε, συνελήφθησαν την παραμονή πρωτοχρονιάς του 7 προς το 8 και καταδικάστηκαν σε, με βαριές ποινές ή αν θέλετε δύο χρόνια και τρεις μήνες και ε, αντίστοιχε ε, ποινές. Είναι, πρόκειται για Ιταλούς που αποδείχθηκε ότι είχαν σχέσεις με την Καμόρα. Πώς το καταφέραμε? Σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Μαφία, όχι ευχαριστώ. Οργανώσαμε λοιπόν ε, και συνεντεύξη που είχαμε μεγάλη απήχηση και έκτοτε η συνεργασία μας εντατικοποιήθηκε περαιτέρω, γιατί πραγματικά ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Για πρώτη φορά εκτός της Ιταλίας αυτή η μορφή συνεργασίας ευωδόθηκε και κατορθώσαμε να συλλάβουμε δράστες της μαφίας. Τώρα, πολύ σύντομα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή, μας, στη διάθεσή μου. Στα πέντε χρόνια αυτή της συνεργασίας οργανώσαμε 50 εκδηλώσεις στο Βερολίνο, Ρομπέρτο Σαβιάνο, Πετραρέσκι, Γιούργεν Ρότ, Κλάουδιο Λακάμερα, Φραντσέσκο Φοτζόνε και με πάρα πολλούς άλλους, με τον Τζοβάνι Ιμπαστάτο, με τον Μικέλε Κόρτο, Ροζάριο Κροτσέτα, δεν ξέρω αν έχει έρθει, νομίζω δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτά που βλέπετε είναι οι προσκλήσεις που απευθύναμε ε, ε, υπάρχει και μία άλλη πρωτοβουλία, η Φλερ. Νομίζω κάποιο που θα ακολουθήσει ο μιλητή θα μιλήσει επ' αυτής. Οι επιτυχίε μα, οι εξή στην Γερμανία αλλά και εκτός αυτής ε, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε όπως σας είπα πρωτοβουλίες να συνενώσουμε ομάδες ε, συμφερόντων κατά της Ιταλίας και μέσα από την αστυνομία όλους αυτούς να τους εντάξουμε σε ένα δίκτυο προστασίας. Το βασικότερο θέμα που μας απασχόλησε είναι πώς είναι δυνατόν η κοινωνία των πολιτών να στηρίξει την αντιμετώπιση της μαφίας. Η αξία της νομιμότητας μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την μαφία, το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα. Mafia Free λέγεται αυτή η πρωτοβουλία. Απευθυνθήκαμε στο Ιταλικό Προξενείο, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα, στους πολιτικούς, στις οικονομικές ενώσεις, ε, στους επιχειρηματίες, ε, στο Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και σε πάρα πολλούς άλλους. Έτσι λοιπόν ε, καταλήξαμε τελικά ε, να οργανώσουμε, όπως σας είπα, πάρα πάρα πολλούς. Τώρα ε, θα συντομεύσω λιγάκι την ομιλία μου. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω το εξή. Η Ντραγκέτα βέβαια τα παρακολούθησε όλα αυτά. Ε, είχαμε μια παρακολούθηση, τηλεφωνική παρακολούθηση, από το Ρέτζο Καλάμπρια ε, μέσω Ιταλής. Οι Ιταλοί μας την παρέπεμψαν. Και εκεί τι λέγανε οι, τα μέλη της Δραγκέντα. Ε, καλύτερα να το αποφεύγουμε το Βερολίνο γιατί εκεί καίει, ε, το έδαφος καίει. Αυτά λέγανε στην Δραγκέντα και αυτό μας χαροποίησε πάρα πολύ. Τελειώντας λοιπόν θα πω και εγώ μαφία, επιθυμείτε μαφία, όχι ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Σίγουρα θα υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά. Με τι ερωτήσει που θα εκτεθούν από του συναδέλφου, ε, τώρα θέλω να δώσω λόγο στον κύριο Λιβυρολό, ο οποίος εκπροσωπεί τη ΦΛΕΡ και θα μα παρουσιάσει την άποψή του σχετικά με την πρόληψη Πώ μπορεί να συνεισφέρει η κοινωνία των πολιτών στον τομέα τη πρόληψη. Παρακαλώ, Λιβιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι πρόεδρος της ε, Γης του Πυρός, Τέρα ε, Τελφόκο. Πρόκειται για μια ενώση η οποία ε, μαζί με τη Λίμπερα δημιουργήσε τη Φλερ. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οργάνωση που είναι υπέρ της ελευθερίας, της νομότητας και των δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Και όπως είπε και ο πρόεδρος της Λίμπερα χτες, γεννείται η οργάνωση αυτή από την πρόκληση να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε την εμπειρία της Λίμπερα και σε, ευρωπαϊκό επίπεδο και να ε, ασχοληθούμε με την καταπολέμηση της ε, μαφίας ε, σε κοινωνικό επίπεδο. Και το είπε ο προηγούμενος ομιλητής, πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδης η συνεργασία μεταξύ όσων ασχολούνται με την καταπολέμηση της μαφίας σε διάφορα επίπεδα. Και είναι απαραίτητο για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα το έργο των διοκτικών αρχών του κράτους ε, και των δικαστικών αρχών, αλλά να είναι απαραίτητο να γίνει και μια πολιτιστική δουλειά η μαφία δεν ε, μπορεί να ιτηθεί αποκλειστικά μόνο με τις συλλήψεις που είναι απαραίτητες, αλλά πρέπει να ξεριζώσουμε ε, αυτό το κακό από την κοινωνία και από όλα αυτά τις προκλήσεις γεννήθηκε η Λίμπερα σήμερα ε, αποτελείται από 1600 πραγματικότητες σε όλη την Ιταλία σήμερα η Φλέρς αυτά τα τέσσερα χρόνια μπόρεσε να μεδοποιήσει πάνω από 40 οργανώσεις από 30 χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο από τον Κάφκαζο, από τις χώρες της Μεσογείου κτλ. Η Φλερ εργάζεται επί τριών θεμάτων. Καταρχήν για την πολιτιστική πρόκληση. Πολύ συχνά η ε, μαφία θεωρούταν στην Ευρώπη ως ένα περιφερειακό φαινόμενο, ένα ιταλικό φαινόμενο. Για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση, ε, ουσιαστικά ε, μιλούσαμε για τη μαφία της Κομπλέτ και της Λουφαπάρα, δηλαδή αναφερόταν μόνο στην Ιταλία. Όμως οι, οι τελευταίες έρευνες μας έδειξαν πως το φαινόμενο της ε, μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι όλο ένα και πιο διεθνές φαινόμενο. Υπάρχουν ε, συνεχώς αποδείξεις ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι διεθνικό έγκλημα. Έτσι λοιπόν αν υπάρχει διεθνικό έγκλημα, αν υπάρχει ε, μια κοινωνική δύναμη κατά της μαφίας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το πολιτιστικό έργο και η Ευρώπη των ενεργών πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών να δείξει ότι είναι δυνατό να αναχαιτιστεί το οργανωμένο έγκλημα, να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα μέσω του κοινωνικού έργου. Έτσι λοιπόν αναζητήσαμε σε όλη την Ευρώπη οργανώσεις που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα αλλά όχι αποκλειστικά με τη μαφία. Και το παράδειγμα του Βερολίνου είναι ένα μόνο παράδειγμα όμως. Ε, στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές εμπειρίες οργανώσεων που συνεργάζονται μαζί μας στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές οργανώσεις που ασχολούνται παραδείγματος χάρη ή με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και επομένως και με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί όπου λείπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολύ συχνά έχουμε ισχυρή παρουσία του οργανωμένου εγκλήματο. Χτε ακούσαμε το παράδειγμα τη οικομαφία ή τη εμπορία ανθρώπων. Είναι δύο πολύ ισχυρά παραδείγματα και στην Ιταλία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια καταπολέμηση και σε κοινωνικό επίπεδο. Και η Λαγκαμπιέντε καταπολεμά την οικολογική μαφία, αλλά Έχουμε ολοένα και πιο συχνέ έρευνε στο θέμα του οργανωμένου εγκλήματο που σχετίζεται με τη διακίνηση των αποβλήτων και φαίνεται ότι από την Ιταλία αρχίζουν να γίνονται κάποια πράγματα, όμω στη συνέχεια αναπτύσσονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όπω παραδείγματο χάρη, ε, έχουμε στην Ρουμανία κάποιε τοποθεσίε αποθήκευση. Και αυτό ένα παράδειγμα. Κατά τα λοιπά, έχουμε και το δίκτυο των ε, συγγενών των θυμάτων. Προσπαθήσαμε να βρούμε τους ανθρώπους αυτούς στην Ευρώπη και προσπαθούσαμε και εδώ να δημιουργήσουμε ένα μικρό δίκτυο το οποίο μεγαλώνει. Θα αναφέρω δύο συγγενείς, ε, την κυρία Τζίντιτς και τον Ηλία που είναι αδερφός ε, ε, του συγγράφου που δολοφονήθηκε στη Ρωσία πριν λίγα χρόνια. Έτσι λοιπόν, ε, όπως ε, είπε πολύ καλά χτες ε, και ο κύριος Λουίτζι Τσότη, πολύ συχνά οι συγγενείς των θυμάτων, αφού έχει τελειώσει το πένθος τους, πολύ συχνά εγκαταλείπονται μόνοι. Στην Ιταλία κάτι τέτοιο δεν γίνεται πλέον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις μεγάλων μικρών δραμάτων και πολύ συχνά εγκαταλείπονται μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί, είτε γιατί το κράτος δεν τους στηρίζει, γιατί δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών να τους στηρίξει. Και έχουμε και το, ε, δουλειά επί της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, το έργο επί τη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αυτέ οι εργασίε ξεκίνησαν όταν ο κ. Φρατιμή, δηλαδή ήταν Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχίσαμε να τονίσουμε πόσο απαραίτητο είναι να έχουμε κοινοτική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την κατάσχεση, αλλά και τη κοινωνική χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει ο νόμος 109 του 2006 που προβλέπει την κοινωνική χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί από την μαφία. Έτσι λοιπόν, ε, ε, το κράτος κατάσχει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από τους μαφιόζους και ε, χάρη σε αυτό το νόμο στην Ιταλία υπάρχει δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία υπέρ της κοινωνίας. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήταν σημαντικό να εξάγουμε αυτή την εμπειρία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα ε, έχει και καταρχήν συμβολικό χαρακτήρα κάτι τέτοιο. Μία από τις πιο μεγάλες εξουσίες που έχει η μαφία είναι να μπορέσουν να κυριαρχήσουν οι μαφιώσεις στην οικονομία δυστυχώς αυτή η οικονομία ε, έχει κάποια εξουσία και σε κάποιες περιοχές, κυρίως στην Νότια Ιταλία, η μαφία είναι η μόνη που δίνει δουλειά. Και το να δίνουμε δουλειά σήμερα σημαίνει να δίνουμε αξιοπρέπεια σε ένα άτομο και σε αυτά τα εδάφη έχουν δημιουργηθεί κάποιες κοπερατίβες από νέους οι οποίοι έχουν ε, αποδώσει στη συλλογικότητα ένα παρουσιακό στοιχείο που μέχρι τα τέλη της διαδικασίας ε, ήταν υπό την κατοχή των μαφιόζων. Τι σημαίνει αυτό, ότι η οικογένεια ε, αυτού του ανθρώπου που είναι και στο οργανωμένο έγκλημα είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στους ανθρώπους που εργάζονταν εκεί. Όμως αυτή η νομοθεσία ουσιαστικά αποκαθιστά την αξιοπρέπεια σε σχέση με την χρήση αυτών των αγαθών. Έχουμε τα προϊόντα της Λιμπερατέρα, της ελεύθερης γης όπως ε, είπαμε χτες, είναι προϊόντα που βρίσκονται σε όλη την Ιταλία και αρχίζουν να και στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Αφενό, έχουμε μια ωραία ιστορία. Υπάρχει δυνατότητα να πούμε ότι για του νέου μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία με καθαρή οικονομία σε τόπου όπου πρώτα είχαμε ε, οικονομία που απασχολούνταν οι μαφιόζοι. Ε, και κατά τα λοιπά έχουμε και μια οικονομική αξία γιατί έχουμε αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο σούπερ μάρκετ και όχι μόνο και αυτό μας δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε καθαρές επιχειρήσεις. Αυτή την πρόκληση εμείς την αντιμετωπίσαμε, αρχίσαμε να εργαζόμαστε με την Επιτροπή για την οδηγία για την κατάσχεση όμως όπως είπαμε και χτες δεν προβλέπεται από την οδηγία αυτή η κοινωνική χρήση των περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει ένα, υπήρξε ένα άνοιγμα από την πλευρά της Επιτρόπου τους προηγούμενους ε, μήνες και Φλέρ και Λιμπερ οργάνωσαν με επίσκεψη της Επιτρόπου Μάλτστρομ ε, σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί στην Ιταλία. Έγινε μια επίσκεψη στην Απουλία όπου είναι πολύ ισχυρό το σύστημα και μιλώ για σύστημα γιατί εκ νέου στην Ιταλία αυτά που έχουν κατασχεθεί, δυνάμει τη νομοθεσία, λειτουργούν εκεί όπου υπάρχει πραγματική συνεργασία με πολιτική κοινωνία ε, των δικαστικών και των αστυνομικών αρχών ε, και του κράτους. Δηλαδή αυτό είναι ένα σύστημα που θέλουμε να εξάγουμε προς την Ευρώπη. Δεν μιλάμε μόνο για την κοινωνική χρήση, αλλά μιλάμε για ε, κάποια δημιουργία θέσεων εργασίας. Έτσι λοιπόν ε, θα ήταν ε, μια δυνατότητα να δείξουμε ότι υπάρχει Ευρώπη των πολιτών αν υιοθετούσε με αυτό το παράδειγμα. Η ΦΛΕΡ είναι μια οργάνωση που αποτελείται κυρίως από τους νέους και θέλει να οικοδομήσει όχι μόνο μια Ευρώπη που θα αποτελείται από νόμους, αλλά και από συγκεκριμένα δικαιώματα και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα με αυτόν τον τρόπο ε, γίνεται και μιλώντας ε, και όχι μόνο για ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και για δικαιώματα του πολίτη. Και θα κλείσω τώρα εδώ με το εξής. Ε, πρέπει να αναφέρω και μια άλλη πρόκληση σήμερα δυστυχώς δεν ε, υπάρχουν ε, οικονομικά και χρηματοπιστωτικά μέσα που να υποστηρίζουν δίκτυα όπως το δικό μας αυτό, γιατί φυσικά είναι μακρύ το έργο. Η Κομισιόν αρχίζει μαζί μας να εξετάζει το θέμα του οργανωμένου κλίματος. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο χρόνια δημιούργησε μια πλατφόρμα που λέγεται ε, πλατφόρμα για ε, την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Έτσι λοιπόν, εκεί ε, συνεδριάζουν κάποιοι αρμόδιοι για να μιλήσουν για το ζήτημα αυτό, για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Εκεί υπήρξαν και κάποιες εμπειρίες της κοινωνίας των πολιτών, εκεί συμμετέχουν και η Λίμπερα και η Φλερ, έχουν... Ε, συνεργαστεί με την Κομισιόν σε αυτό το θέμα σε σχέση με τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία και την ιταλική εμπειρία. Έχει γίνει μια δουλειά ευαισθητοποίηση αλλά και μια δουλειά οικονομικού χαρακτήρα. Σήμερα δεν υπάρχουν κάποιοι διαγωνισμοί που να ευνοούν τέτοιε εμπειρίε που να ευνοούν την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο σε κοινωνικό επίπεδο. Υπάρχουν μορφέ χρηματοδότηση για τι διοκτικέ ορχέ καταρχήν, που ασχολούνται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. όμω θα ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόκληση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αρχίζει να χρηματοδοτεί και τέτοια κοινωνικά δίκτυα. Θα ήταν ένα τρόπο να δώσει αξιοπρέπεια στα δίκτυα αυτά και να του αναγνωρίσει ένα πραγματικό ρόλο. Και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, τον κύριο Αλότο και τώρα ε, θα υποβληθούν ερωτήσεις ε, και μετά θα έχουν δυνατότητα οι ομιλητές να απαντήσουν. Θα ήθελα να μην μακρηγορείτε ή δυνατόν να υποβάλλετε απευθεία την ερώτηση έτσι ώστε οι προσκεκλημένοι μας να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Ο κύριος Γιακολίνο, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε τους ε, δύο εισηγητές, ε, τον κύριο Φίνγκια, ε, κυρίως που είναι στην αστυνομία 43 ολόκληρα χρόνια. Μας παρουσίασε λοιπόν το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε επίπεδο πρόληψης, αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος στη Γερμανία. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ και να ρωτήσω σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα και τα μέσα, τα νομικά μέσα που έχει κανείς για να τα αντιμετωπίσει. Εμείς έχουμε κάνει την εξής εμπειρία. μετά το Ντούισμπουργκ της ε, Γερμανίας ε, πράγματι προέκυψε κάποια ευαισθητοποίηση και στα άλλα κράτη-μέλη. Γιατί εκεί διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις τουλάχιστον όσον αφορά την ε, συνεργασία των αστυνομικών αρχών. Αυτή η πρωτοβουλία μαφία όχι ευχαριστώ. Αυτή πράγματι ήταν μια πολύ αποτελεσματική πράξη και γι' αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την ευαισθησία που επιδείξατε. Κατά τα άλλα, ε, θέλω να σας πω ότι ε, ε, θα προσπαθήσουμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε αυτά που προβλέπονται στην Ιταλία και στην Ισπανία αν θέλετε να μεταφερθούν και σε ολόκληρη την Ευρώπη έτσι ώστε να υπάρχει ή δυνατόν κάποια ομοιογένεια σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιακολίνο εκ μέρου ε, της ΑΛΔΕ των Φιλελευθέρων ο κύριος ε, Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ κύριε Φίγκερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε υποθέτω από το Βερολίνο. Είναι μακριά. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Γιατί εδώ δεν ε, κάνουμε έρευνα για την μαφία. Μία χώρα από τις 27 ίσως να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτήν φυσικά. Πολύ χαιρόμαστε που ακούμε ότι δεν υπάρχουν πολλές δραστηριότητες της μαφίας ή της Καμόρας στο Βερολίνο. Αλλά για τους Ρώσους, για τους Κινέζους, για τους Ανατολικοευρωπαϊκούς ή για άλλου είδους οργανωμένο έγκλημα έχετε να μας πείτε κάτι γιατί εμείς και γι' αυτό θέλουμε να ξέρουμε, γιατί εμεί ερευνούμε για ολόκληρη την Ένωση. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Η μαφία μπορεί να έχει δύναμη στην Ιταλία. Εσείς είσαστε σε μια από τις πιο σημαντικές πρωτεύουσε της Ευρώπης. Σίγουρα έχετε πάρα πολλά πράγματα να μας πείτε για λαθρεμπόριο, ναρκωτικών, όπλων και για ένα σωρό άλλες δραστηριότητες. Αν έχετε χρόνο λοιπόν θα μπορούσατε να επεκταθείτε λιγάκι και προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για σας, εγώ δεν είχα ακούσει αυτή την περίπτωση. Με το iPad μου εδώ πέρα άρχισα να το ψάχνω, αλλά εσείς έχετε κάποια ιστοσελίδα για να διαβάσω γι' αυτό, γιατί εγώ ειλικρινά για την δικιά σας την οργάνωση, την Terra de la Fuoco, δεν βρήκα πολλά πράγματα. Βλέπετε, εγώ είμαι στα East Midlands, στην Αγγλία, που φυσικά δεν συγκρίνονται, αλλά θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για σας και θα ήθελα να μου πείτε πού μπορώ να τις βρω. Ματιέ, η κυρία Ματιέ για δύο λεπτά από το ΕΛΚ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Φίγκερ, λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ γιατί άργησα να φτάσω και δεν άκουσα ολόκληρη την παρουσίασή σας, η οποία δίχως άλλο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλιώς δεν θα ήσασταν και εδώ. Δεν θα Σα ρωτήσω πολλά γιατί ξέρω για την μαφία, αλλά κύριε Λότε σα άκουσα την παρουσίασή σας, πολύ ενδιαφέρουσα και για την Ιταλία βέβαια, αλλά έχω δύο ερωτήσεις. Υπήρξε, υπάρχουν επιπτώσεις από την οικονομική κρίση την τόσο σοβαρή που διανύουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στην Ιταλία. Υπάρχουν επιπτώσεις στη δραστηριότητα της μαφίας. Εσείς λέτε ότι οι μαφιόζοι βρίσκουν δουλειά στους ε, απλούς πολίτες και γι' αυτό και έχουν τη συμπαθιά τους μερικές φορές. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ενεργεία και στην Ιταλία και αλλού. Λοιπόν, ρωτάω, υπάρχουν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της μαφία από την κρίση αυτή. Δεύτερον, μπορεί να μην είναι politically correct, να μην είναι ορθή πολιτικά. Θα την κάνω όμως. Το Βατικανό παίζει ρόλο στην μαφία. Ελπίζω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Ευχαριστώ. Και χωρίς να χρησιμοποιήσετε ξυλίνη γλώσσα. Ευχαριστούμε. Γκουε, ο κύριος Άντεργκαρτ. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι πρώτα τον κύριο Φίγκερ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι απ' έξω μας έρχονται όλα. Εύκολο είναι αυτό. Για τη Δανία δεν θα έλεγα το ίδιο, γιατί η πιο σημαντική απειλή για τη δημοκρατία έρχεται από δανέζικες εγκληματικές οργανώσεις, που έχουν βέβαια διεθνή δίκτυα. Όμως, εμείς οι ίδιοι βρίσκουμε τη δικιά μας εγκληματικότητα. Δεν πρέπει δηλαδή κάθε φορά να καταδεικνύουμε τους άλλους και να λέμε ότι οι άλλοι φταίνε για τη δικιά μας εγκληματικότητα. Δεν είναι πάντα εισαγόμενοι. Τώρα μας ε, μιλήσατε για το γερμανικό οργανωμένο έγκλημα. Οι bikers, οι bendidos, οι black angels κλπ. Όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το λαθρεμπόδιο ναρκωτικών που απειλούν τον κόσμο, που τον σκοτώνουν ή που άλλοι σκοτώνονται. Πώς αντιδράει η Γερμανία. Οι hedge Angels έχουν βέβαια απαγορευτεί. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες ε, πληροφορίες για το υπόβαθρο. Εσείς στη Γερμανία γιατί έχετε ακολουθήσει αυτή την πολιτική και έχει φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σελήνο για δύο λεπτά. κύριε Πορσελίνο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φίγκερ για αυτά που είπε στην αρχή και υπενθύμησε την 20η επέτειο από την σφαγή στο Παλέρμο. Οι ερωτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι έβαλαν βέβαια το όλο θέμα σε ε, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής μόνο η Ιταλική μαφία, δηλαδή πιο συγκεκριμένα η Ντράγκητα, αλλά ας πούμε η Ιταλία, η μαφία είναι εκείνη που υπάρχει στην Ιταλία, μόνο αυτή. Δεν αναφέρομαι στη Ρωσική, την Κινέζικη ή σε άλλες μαφίες. Εγώ, εμένα με ενδιαφέρει η τοπική εγκληματικότητα που έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει δίκτυα με την Ντράγκητα και να οικειοποιείται το μήνυμα που θέλει να περάσει η Ντράγκετα. Ερωτώ συγκεκριμένα, η μαφία στη Γερμανία είναι εισαγόμενη, μόνο εισαγόμενη ή μήπως υπάρχει και ε, τοπική εγκληματικότητα η οποία απλά οικειοποιείται τα μηνύματα της Ιταλικής εγκληματικότητας. Και επίσης ε, θα ήθελα να πω στον Ολιβιέρο που τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η δραστηριότητα την οποία αναπτύσσεται την ε, εκτιμώ ιδιαίτερα. Και αυτό διότι όταν ε, παρουσιάστηκε η Λίμπερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν νομίζω το 98 τότε. Θυμάμαι τους ε, συναδέλφους από τότε. Εντάξει, εγώ τότε δεν ήμουν ευρωβουλευτής. Πάντως οι ίδιοι είπαν ότι ε, θαυμάζουν αυτή την πρωτοβουλία στην Ιταλία που αναπτύσσει αυτή την δραστηριότητα. Εκτιμώ λοιπόν ιδιαίτερα τη δουλειά σας. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα προς τα μπρος και είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν και άλλα. Επιτρέψτε μου βέβαια λίγο έτσι κάπως να αμφισβητήσω αυτό που είπες ότι στην ε, Νότια Ιταλία η μαφία είναι εκείνη η μόνη που είναι εργοδότης και που δίνει δουλειά. Δεν είναι αλήθεια. Δεν δίνουν παίρνουν δουλειά, την παίρνουν από ένα τομέα και την δίνουν σε άλλο. Και αυτό καταστρέφει την οικονομία. Είναι λοιπόν χειρότερη η κατάσταση αντί ε, να είναι καλύτερη όπως ε, την παρουσίασε εσύ. Απλά έτσι αυτή τη μικρή αμφισβήτηση ήθελα να κάνω. Βάντεν Χόλσεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που ακούσαμε γιατί νομίζω ότι όλα αυτά ενείχαν την ευρωπαϊκή διάσταση. Σήμερα ακούσαμε παραδείγματα από την Ιταλία, Ιταλικά δίκτυα. Πιστεύω όμως ότι από αυτά μπορεί κανείς να συνάγει γενικότερα συμπεράσματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό που είπε ο κύριος Φίγκε, ότι υπάρχει μια άμεση διασύνδεση με την κοινωνική κατάσταση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους καταστάσεις προκύπτουν συχνότατα λόγω λόγω ένδυας. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά σοβαρά. Όποιος δεν επενδύει σε κοινωνική υποδομή, μετά εκ των υστέρων καλείται να πληρώσει ε, τεράστια κονδύλια για την δημιουργία δικτύων ασφαλείας. Η κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το σκεφτούμε. Τι σημαίνει ακριβώς στην Ευρώπη πολιτισμός της νομιμότητας, νοτροπία νομιμότητας. Το κράτος δικαίου, η υπεροχή του κράτους δικαίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και από ό,τι φαίνεται ε, καλείται κανείς να το διεκδικεί συνεχώς. Αυτό παίζει ρόλο όχι ε, στην διαφώτιση αλλά και στην πρόληψη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ε, οι οποίοι πιστεύουν στο κράτος δικαίου και αυτοί δεν είναι ευεπίφοροι για ε, τρομοκρατικές ε, δραστηριότητες, για την εμπλοκή τους σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Και προς τον κύριο Φίγκε, ερωτώ, εσείς γνωρίζετε μόνο το μοντέλο του Βερολίνου ή μήπως ξέρετε να υπάρχουν και άλλα συγκρίσιμα μοντέλα σε άλλες γερμανικές πόλεις. Και ρωτώ αυτό που ρώτησε και ο, ο Βρετανός συνάδελφος καταφέρατε να απευθυνθείτε και σε άλλες κοινότητες, γιατί δεν έχουμε μόνο την Ιταλική μαφία, είναι λιγάκι άδικο να μιλάμε συνεχώς ε, για την Ιταλία. Ε, το φαινόμενο θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ευρωπαϊκό. Και άλλη μία ερώτηση προς τον κύριο Αλότο. Κύριε Αλότο, Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εκπονηθούν και άλλα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν τις δικές σας τις δραστηριότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει η Πρόεδρος, ε, δύο λεπτά ε, στον κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνο απόλυτα με τον κύριο Σόντεγαρτ για το ότι ο καθένα στη χώρα μας έχουμε τη δικιά μας εγκληματική οργάνωση, αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει διασυνοριακό έγκλημα. Δανία, Σουηδία, έχουμε μια γέφυρα μεταξύ μας. Αφού τη χτίσαμε αυτή τη γέφυρα, άλλαξε το περιβάλλον. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Πάντα ήμουνα υπέρ της γέφυρας αυτής, παρά το γεγονό ότι πολλοί πολίτε έλεγαν τότε ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα, γιατί από την Κοπεχάγη θα πάει στη Σουηδία στο Μάλμε η εγκληματικότητα, είτε πρόκειται για τους μπαντίδους, είτε για την Black Cobra, είτε για οποιαδήποτε άλλη εγκληματική οργάνωση. Ή ανάποδα βέβαια. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί εννοείται ότι είναι πολύ βασικό στοιχείο τα ανοιχτά σύνορα, μόνο που γίνεται κατά χρυσή τους από τις εγκληματικές συμμορίες. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν κάτι για τους bikers. Στην αρχή για τους bikers. Στην αρχή αυτή, έτσι σκληρή, τους αναγνωρίζει κανείς εύκολα και από το εξωτερικό τους, την εξωτερική τους εμφάνιση, είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Λοιπόν, κύριε Φίγκερ, εσείς πώς τους αντιμετωπίζετε στη Γερμανία. Ξέρω ότι υπάρχουν και στη Γερμανία. Εσείς πώς ε, χειρίζεστε την περίπτωσή τους δίνεται την εντύπωση, μάλλον δίνουν την εντύπωση ότι αποτελούν μέρος της κοινωνίας. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Γιατί πώς θα προστατεύσουμε τους μαγαζάτορες, ε, τον κόσμο, όταν ε, αυτοί πάνε και λένε στους μαγαζάτορες, για παράδειγμα, ότι εμείς θα σας προστατεύσουμε από άλλες συμμορίες. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στους προσκεκλεισμένους μας, θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φίνκερ. Αν παραδεχτούμε την αναγκαιότητα να θέσουμε σε ένα πλαίσιο ε, τις επιχειρηματικές σας δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο των εργασιών σας, βάση και τις συνειδητοποίησης ότι η Ιταλική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος είναι η πιο πλήρης και η πιο ειδική. Εσείς, τι δυσκολίες συναντάτε σε ό,τι αφορά τις έρευνες όταν ε, έρχεστε αντιμετωπώς με μια σειρά δικτύων ε, εγκληματικών συστημάτων και αν ε, δούμε και τι συνέβη στο Duisburg. Αν θεωρείτε ότι το αδίκημα της σύστασης μιας μαφιόζικης συμμορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της μαφίας, δηλαδή να έχουμε μια συγκεκριμένη κατηγορία αδικήματος και να ρωτήσω και τον άλλο καλεσμένο μας ε, αν ε, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ΦΛΕΡ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχατε τη δυνατότητα να συναντήσετε κάποιες πραγματικότητες παρόμοιες με τις δικές σας στην Ευρώπη και ποιες δραστηριότητες υλοποιήσατε ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε και υπάρχουν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιες πραγματικότητες ε, που να συνάδουν με τη λιτανική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ε, δίνω πέντε λεπτά στους δύο προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Okay. Um... Ich äh, will zunächst Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας επισημάνω ότι σήμερα εγώ ασχολούμαι με την ε, πρόληψη, αλλά σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Ε, και εγώ δεν εκλήθην εδώ για να σας μιλήσω γενικότερα για το διεθνές έγκλημα. Δεν μου το είχατε πει, αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν και άλλα ε, μοντέλα πρόληψης στην Ευρώπη, όμως ε, δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα. Αυτή που είναι πραγματικά ανεπτυγμένη είναι η συνεργασία που έχουμε στο Βερολίνο και η ε, πολυτομεακή ομάδα εργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ε, οργανωμένο έγκλημα το 2009 μας κατέταξε στον κατάλογο των best practices. Είμαστε λοιπόν σε αυτό τον κατάλογο και προσπαθούμε τα δικά μας τα μοντέλα να τα ε, διαδώσουμε και σε άλλα κράτη. Αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν είναι η συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών και των αστυνομικών αρχών και οι δύο από κοινού μπορούν να επιτύχουν πάρα πολλά. Όσον αφορά στην πρόληψη, αυτό που ενδιαφέρει είναι η αντιμετώπιση κινδύνων με βάση τον νόμο και βεβαίως η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο σύνολό του. Όλα αυτά ξεκινούν από την παιδική ηλικία, ε, πάνε την σχολική εκπαίδευση, σε κατάρτιση, μαθητεία, οικογένεια. Ε, όλοι αυτοί οι τομείς ε, καλούνται να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό λοιπόν και σας ε, επισήμανα την σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να αναφερθώ περισσότερο στη Γερμανία. Εμείς έχουμε ιεραρχήσει τις εθνότητες. Στη Γερμανία έχουμε πάνω από 60 εθνοτικές ομάδες που εμπλέκονται σε οργανωμένο έγκλημα. Η Ιταλική τώρα κοινότητα, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά οι μαφίες που έρχονται κυρίως από την Ιταλία βρίσκονται στην τρίτη θέση. Πρώτη, ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι, οι Γερμανοί οι Γερμανοί, όπως και στην Δανία. Οι Γερμανοί είναι οι ε, πολίτες εκείνοι οι οποίοι στη Γερμανία έχουν ενταχθεί στο οργανωμένο έγκλημα. Αλλά και αυτοί οι Γερμανοί αναπτύσσουν κυρίως διεθνείς δραστηριότητες. Η εμπειρία της, της δικής μας της αστυνομικής αρχής είναι ότι περίπου 80% των διαπρατώμενων εγκλημάτων έχουν διεθνή διάσταση. Εντάσσονται δηλαδή στο οργανωμένο έγκλημα, στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Και όταν λέω για τον 80% αυτών των εγκλημάτων, προφανώς δεν αναφέρουμε μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Καναδά, Αυστραλία, σε όλες τις υπήρους. Προφανώς και την Κίνα αναφέρουμε και στο σύνολο του ασιατικού χώρου. Τώρα, όσον αφορά στο ερώτημα για την στοχευμένη αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών εγκληματικότητας, όπως αυτή η εγκληματικότητα των rockers. Πριν από λίγες μόνο ημέρες ε, μίλησα με την ε, αρμόδια αρχή στο Βερολίνο που ασχολείται με τους Hells Angels. Ε, την εγκληματικότητα των rockers την αντιμετωπίζουμε πολύ αυστηρά γιατί πρόκειται για διεθνώς οργανωμένη εγκληματικότητα. Είναι άτομα τα οποία ασκούν βία με ιδιαίτερο τρόπο και έχουν μάλιστα και πολύ καλή διεθνή δικτύωση. Αυτή είναι πολύ καλά οργανωμένη ε, στα ναρκωτικά αλλά και στα ε, όπλα και στην εξαναγκαστική πορνεία. Άρα δηλαδή εμπλέκονται και σε θέματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Και εδώ ε, πρέπει να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δηλαδή αποτροπή κινδύνου αλλά και ποινική δίωξη. Εγώ έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου για τη διαφοροποίηση αυτών των bikers γιατί εμείς ε, ως αστυνομία και ως κράτος πρέπει να έχουμε διαφοροποιημένη προσέγγιση, να προχωράμε συνετά. Δεν είναι το ότι οι bikers ε, είναι όλοι εγκληματίε και εγώ έχω μοτοσυκλέτα. Και εγώ μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ. Δεν είναι όλοι οι μοτοσυκλετιστές εγκληματίε. Εμάς μας ενδιαφέρει να επιλέξουμε τους εγκληματίες, μοτοσυκλετιστές, ε, αυτούς ε, που νιώθουν έτσι λίγο easy rider. Αυτοί όμως, πολλοί εξ αυτών, είναι εγκληματίες, εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους. Δεν μιλάμε συνολικά για τους μοτοσυκλετιστές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προχωράμε διαφοροποιημένα. Δεύτερη παρατήρηση. Υπάρχει ε, το εξή μοντέλο, το οποίο και σας ε, παρουσίασα. Είναι ένα μοντέλο που προέρχεται από την Ιταλία, έχει φτάσει στο Ντουίσμπουργκ, επεκτείνεται στους Άραβες, στους Τούρκους, Έχουμε τους ε, Σίντι και τους ε, Ρωμά. Αυτούς τους ε, εντάσσουμε σε κύκλους επικοινωνίας, σε συζητήσεις με μας. Συζητάμε και εκεί μορφές εγκληματικότητας μονομένων μελών των Ρουμάνων και των Πολωνών Σίντι και Ρωμά. Θέλω να πω ότι επεκτηνόμετα και σε άλλες εθνικότητες και εθνοτικές ομάδες. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η Ιταλική νομοθεσία είναι πολύ πιο προχωρημένη από τη Γερμανική και από πολλές άλλες ε, νομολογίες και νομοθεσίες άλλων κρατών μελών. Γι' αυτό και εμείς επιθυμούμε ότι είναι καλό και σωστό να το εισάγουμε στην Ευρώπη ή αν θέλετε να το εξάγει η Ιταλία έτσι ώστε σε τελική ανάλυση να κατορθώσουμε στην Ευρώπη την, να επιτύχουμε την εναρμόνιση των νομοθεσιών και σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών πολύ συνετά να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά εκείνες τις ομάδες οι οποίες διαπράττουν κοινωνικό κακό. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Αλότο για πέντε λεπτά. Ναι, σας ευχαριστώ για τις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχήν για την ερώτηση του κυρίου Νιουτοντάν για την οργανωσή μας ε, και στο Τωρίνο teradelfoco.org ε, είναι η ιστοσελίδα. Εμείς εργαζόμαστε πάρα πολύ για τους πρόσφυγες και για τους Ρωμά και για το θέμα της μετανάστευσης και ε, αρχίσαμε να γνωρίζουμε το θέμα του οργανωμένου κλίματος, ε, ξεκινώντας με την ενασχόληση με τους Ρωμά, τους μετανάστες ε, και τους πρόσφυγες και ιδίω στην ε, Βορεια Ιταλία δυστυχώς οι μετανάστες είναι ε, το πρώτο κύκλο μου που πάει να ψαρέψει το οργανωμένο έγκλημα. Καταρχήν γιατί πρόκειται για άτομα που βρίσκονται σε αδύναμη κατάσταση και χρειάζονται εισόδημα και πολύ συχνά και στις χώρες ε, προέλευσης είναι θύματα. Σκεφτείτε την εμπορία ανθρώπων, παραδείγματο χάρη όταν μιλάμε για ανθρώπου που προερχόνται από τη Βορεια Αφρική που πληρώνουν τεράστια ποσά για να φτάσουν στην Ευρώπη αλλά και μόλις φτάσουν πολύ συχνά συχνά είναι θύματα εθνικών κυκλωμάτων, εγκληματικών κυκλωμάτων, γιατί η μικροεγκληματικότητα αυτό χρειάζεται. Και κατόπιν οι άνθρωποι αυτοί εξυπηρετούν το κέρδος των μεγάλων εγκληματιών. Έτσι λοιπόν από εκεί γεννήθηκε η ασχολούμαστε με το οργανωμένο έγκλημα στην Ιταλία, εργαζομένοι στα σχολεία, κάνουμε ένα πολιτιστικό έργο, αλλά και πιο συγκεκριμένα ασχολούμαστε και με τη μετανάστευση. Προσπαθούμε λοιπόν να συνδέσουμε το θέμα των δικαιωμάτων με το θέμα των καθηκόντων. Το δικαίωμα στο στέγη επιτρέπει στους μετανάστες που φτάνουν στην Ιταλία να έχουν μικρότερες πιθανότητες να μπουν σε εγκληματικά κυκλώματα. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ε, σειρά συνδέσεων στην Ευρώπη και από εκεί γεννήθηκε και η εμπειρία του Φλερ. Δεύτερη ερώτηση. Το θέμα της κρίσης η εμπειρία που έχουμε εμεί, θα σα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα σχετικά με την εμπειρία μα. Φυσικά η κρίση αύξησε τη δύναμη του οργανωμένου κλίματο και τη μαφία. Τρία παραδείγματα. Ε, το θέμα τη τώρα κάποια στιγμή που εμεί έχουμε ε, ουσιαστικά ε, να σκεφτούμε τι γίνεται με την οικονομία, με τις πιστώσεις, ε, πόσο, ε, πόσο, πόσο δύσκολη κατάσταση είναι οι επιχειρήσεις για να δανειστούν. Έχουμε κάποιες άλλες εγκληματικές οργανώσεις που δεν έχουν πρόβλημα ρευστότητας και φυσικά οι επιχειρηματίες και όχι μόνο παρουσιάζονται ενώπιον αυτών και ζητούν μια συγκεκριμένη ε, δυνατότητα να έχουν ε, γρήγορα ρευστότητα. Έτσι λοιπόν ε, ε, υπάρχει αυτή η διευκόλυνση από τη μαφία και αυτό είναι ένα θέμα που συμβαίνει στην Ιταλία, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και δυστυχώς όχι μόνο στην Ιταλία και προχτές ε, συμμετείχα σε μια διάσκεψη όπου έχουμε ένα Ινστιτούτο που συνδέεται με τους τοκογλήφους και με τους εκδιασμούς και υπάρχει πολύ μεγάλη σύνδεση ε, με το τι συμβαίνει στην Ιταλία, με τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα δάνεια που παίρνουν τα άτομα και πρέπει να πληρώνουν πολύ ψηλούς τόκους, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλα κεφάλαια προ προέρχονται από την Ιταλία, αλλά πολύ συχνά επενδύονται στο εξωτερικό. Ε, η μαφία λοιπόν δεν πληρώνει την κρίση. Έχουμε δύο αγορές που μας δείχνουν ότι δεν είναι σε κρίση. Τα ναρκωτικά και οι κατασκευές. Η αγορά των ναρκωτικών δημιουργεί τόσο μεγάλη ροή χρημάτων και Έχετε συζητήσει εσείς και για αυτό το θέμα ως ε, Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν σε τέτοιες καταστάσεις ε, συνεχώς χρήματα κυκλοφορούν και ουσιαστικά ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και Έχουμε και άλλα παραδείγματα, όπω το χάρη διακίνηση όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων. Ποτέ δεν υπάρχει κρίση σε αυτού του τομεί. Εκμεταλλεύονται λοιπόν οι μαφιόζοι την κρίση της νομιμότητας. Κύριε Μπορσελίνο, ίσω ε, να μην τα καλά, το θέμα είναι αυτέ οι γκρίζες ε, ζώνες για το Βατικανό και για την Εκκλησία. Είναι σαφές ότι στην Ιταλία έχουν υπάρξει κάποιες εμπειρίες ε, διασύνδεσης της Εκκλησίας του Βατικανού με τη μαφία, αλλά θέλουμε έχουμε και πολύ ισχυρό Βατικανό σε ό,τι αφορά την κοινωνική παρέμβαση. Και κάτι ακόμη, το κράτος ε, του Βατικανού βρίσκεται υπό μία έρευνα αυτές ε, τις μέρες και παρουσιάζεται και στις εφημερίδες, ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Ίσως να μην μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για μαφία, αλλά για οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή υπάρχει σύνδεση του οργανωμένου έγκληματος και του κράτους του Βατικανού γιατί ξέρετε και η ιδιαιτερότητα της ε, μαφίας είναι ακριβώς αυτό. Ναι, υπάρχει διασύνδεση εγκληματικότητας και κράτους. Έτσι λοιπόν, όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει μια εκκλησία που δείχνει ένα πιο κοινωνικό χαρακτήρα και απέναντι σε αυτό. Νομίζω ότι ε, αναφέρθηκε και το παράδειγμα χτες ε, πολύ μικρών ενοριών που απαντούν στο οργανωμένο εγκλήμα. Λοιπόν, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα η Επίτροπο Μάλστρομ και η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ εσωτερικών χρηματοδοτεί προγράμματα καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Πρόκειται ένα, για ένα πρόγραμμα που λέγεται EZEX. Στο εσωτερικό αυτού του προγραμματό με κανένα τρόπο δεν ε, υπάρχουν προγράμματα ειδικά για την κοινωνία των πολιτών. Έτσι λοιπόν, από την ε, πλευρά τη Επιτρόπου και του Γενικού Διευθυντή γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε στη χρηματοδότηση του 2014 να μπει και η χρηματοδότηση Τη της καταπολέμησης του οργανωμένου κλίματος σε κοινωνικό επίπεδο. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με την Αρμόδια και είχαμε και μία επίσκεψη της Επιτρόπου σε αυτή τη γη που έχουμε κατασχέσει προκειμένου να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα και σε πολιτικό επίπεδο βέβαια αυτό θα σημαίνει ότι θα δώσουμε μια αξιοπρέπεια ε, στην κοινωνία των πολιτών που καταπολεμά το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα ήταν λατασμένο να έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, θα ήταν πολύ καλύτερο στο εσωτερικό ε, των κονδυλίων που ε, ήδη αφιερώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του οργανωμένου έγκληματος να έχουμε και αυτή την χρηματοδότηση της κοινωνικής συνιστώσας. Έχουμε και την ερώτηση της κυρίας ε, Αλφάνο. Δύο παράδειγματα θα αναφέρω. Σκέφτομαι το Κωσυφοπαίδιο, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Και συγκεκριμένα το νησί στη Σερβία, όπου υπάρχει μια οργάνωση που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων ε, και προσπαθεί ουσιαστικά να κόψει τις γέφυρες μεταξύ μετανάστευσης και οργανωμένου κλίματος. Στο Μαυροβούνιο έχουμε δύο ενώσεις, μία νέων και μία μη νέων, που ασχολούνται με την ομοποίηση παράνομων εσόδων και με τη σύνδεση μεταξύ αυτής της νομοποίησης παράνομων εισόδων και διαφθοράς. Είναι πραγματικά μια ισχυρή δουλειά κοινωνικού χαρακτήρα και θα ήταν ενδιαφέρον και για την Επιτροπή, δεν ξέρω αν το προβλέπετε στις εργασίες σας, να βρείτε και πραγματικότητες εκτός της Ιταλίας, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ιταλία. Ωραία θα ήταν να μας επισκεφτείτε και σε αυτά τα κατασκευμένα εδάφη ε, για να δείτε τι στην πραγματικότητα συμβαίνει εκεί, για να εντάξουμε και στην οδηγία αυτή την πρόβλεψη για την κοινωνική χρήση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο μίλητες. Την επόμενη εβδομάδα να σας πω ότι δεν ε, ολοκληρώνονται εδώ οι δραστηριότητες της Επιτροπής μας, αλλά συνεχίζονται την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, γιατί θα έχουμε μια αποστολή στη Σερβία. Ίσως λοιπόν να μας δώσετε αυτές τις επαφές, γιατί θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας θα είναι στην Ιταλία τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου με μια συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίστηκε πραγματικά να επισκεφτούμε αυτά τα εδάφη που έχουν κατασκευθεί, που έχουν κατασκευθεί έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εμείς ως ε, Επιτροπή έχουμε σχεδιάσει ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε για να είμαστε χρήσιμοι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη συνεισφορά σας και που ήσασταν τόσο σαφείς και ειλικρινείς στις απαντήσεις σας. Συνεχίζουμε τώρα με την ε, τελευταία ομάδα. Αυτήν, ε, όπως σας είπα, η τελευταία συνεδρίασή μας πριν από τις θερινές διακοπές. Όμως ε, συνεχίζουμε, τη Δευτέρα θα είμαστε στις αποστολή στη Σερβία. Τώρα, οι δύο τελευταίες παρεμβάσεις έχουν να κάνουν ε, με θέματα πάρα πολύ ευαίσθητα, τα οποία συχνά έχουμε συζητήσει. Καταρχήν, έχουμε την διαχείριση στα σοφρονιστικά καταστήματα και τη μορφή εφαρμογή και εκτέλεση των ποινών για τα ε, αδικήματα του οργανωμένου εγκλήματο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ έχουμε καλέσει τον κύριο Καστιλέχο, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της Ισπανικής ε, δίκηση των Φυλακών και κατόπιν έχουμε τον ε, κύριο ε, της υπηρεσία του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πάλι θα δώσουμε 15 λεπτά στους καλεσμένους μας και 2 λεπτά για τους υπόλοιπους συναδέλφους, εισηγητές, συντονιστές και μέλη της Επιτροπής. Έτσι λοιπόν θα δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Καστιγέχο, ο οποίος ε, θα μας παρουσιάσει την άποψή του σε σχέση με τη διαχείριση των σοφρονιστικών καταστημάτων και με τον τρόπο εφαρμογής και εκτέλεσης ε, των ποινών όταν μιλάμε ε, για εγκλήματα, για το οργανωμένο έγκλημα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την δυνατότητα αυτή να συμμετάσχω στην ειδική αυτή επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειλικρινά ευχαριστώ και την Πρόεδρο για την πρόσκλησή της. Θα μιλήσω ισπανικά. Το διασυνοριακό έγκλημα αποτελεί απειλή για την ειρήνη και για την ανάπτυξη, αλλά και για την ίδια την κυριαρχία των εθνών. Αυτά τα είχε πει ο Αντώνη Μαριακώστα, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, της Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του εγκλήματος και των ναρκωτικών. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα που προποθέτει την ε, ύπαρξη εγκληματικών οργανώσεων με συγκεκριμένους κανόνες και με συγκεκριμένους στόχους που μπορεί να είναι πολιτικοί στην περίπτωση της τρομοκρατίας, αν και από την εμπειρία που έχω εγώ όσον αφορά την τρομοκρατία στη χώρα μου, έχουν και μαφιόζικους τρόπους λειτουργίας, αλλά από την άλλη μπορεί να πρόκειται και για στόχους ε, οικονομικού κέρδους απλά. Η οργάνωση Πάντως μεταφέρει αυτούς τους στόχους και σε, όλους τους, σε όλα τα μέλη τα οποία προσχωρούν σιγά σιγά. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εγκληματικέ οργανώσεις, είτε ασχολούνται με την ανατροπή καθεστώτων εξουσίας, είτε πρόκειται ε, για στόχο το κέρδος, είτε για οτιδήποτε άλλο. Στην Ισπανία τώρα πρέπει να σας πω ότι η ποινή φυλάκισης έχει σαν στόχο την ε, μετάνοια του κρατούμενου, αλλά και την αποτροπή άλλων τέτοιων περιπτώσεων. Στόχος μας κυρίως είναι η αποκατάσταση, δηλαδή του κρατούμενου προκειμένου να πετύχουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Τώρα, οι σοφρονιστικοί τρόποι που χρησιμοποιούμε δεν πρόκειται να πετύχουν εάν δεν εφαρμοστούν σωστά για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, το οποίο βέβαια αλλάζει όσο περνά ο καιρός. Οποιοδήποτε σοφρονιστικό σύστημα σε μια δημοκρατική χώρα πρέπει να συνδυάζει τον στόχο της αποκατάστασης του κρατούμενου έτσι ώστε αυτός να μπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία όταν ολοκληρώσει την ποινή του με την επιθυμία να τηρεί το ποινικό δίκαιο. Δηλαδή, η στάση του κράτους απέναντι στον παραβάτη πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών οι οποίοι μπορεί να πληγούν είτε από έναν ενδυνάμει παραβάτη είτε από έναν παραβάτη ο οποίος έχει διεκτήσει την ποινή του. Στην Ισπανία έχουμε τον Οργανικό Σοφρονιστικό Νόμο του 1979. Στο αρχικό του άρθρο δεν αναφερόταν καθόλου όμως στο οργανωμένο έγκλημα. Ούτε ανέφερε ειδικά μέτρα για την ε, μεταχείριση των κρατουμένων οι οποίοι ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση. Στη συνέχεια όμως το 2003 τροποποιήθηκαν ορισμένα άρθρα του ποινικού δικαίου Οπότε εκεί συμπεριλαμβάνονται διάφορα μέτρα που έχουν να κάνουν με το σοφρονιστικό σύστημα. Για παράδειγμα, οι κρατούμενοι εξαιτία συμμετοχής τους σε οργανωμένο έγκλημα συμπεριλαμβάνονται πια. Βέβαια εξαρτάται από το πόσο επικίνδυνοι είναι οι κρατούμενοι αυτοί και ανάλογα εφαρμόζονται και τα σοφρονιστικά μέτρα. Γι' αυτό και υπήρξε ε, μεταρρύθμιση του ποινικού μας δικαίου το 1996. Πρέπει να σας πω τώρα ότι στη χώρα μου υπάρχει ένα ειδικό δικαστήριο που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για να δικάζει τους εγκληματίες από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία με έδρα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και έχει αρμοδιότητα για ολόκληρη τη χώρα. Είναι η Αουδιένθια Nacional. Σε σχέση τώρα με την έκτηση ποινής, Υπάρχει επίσης ένα ειδικό δικαστήριο το οποίο ελέγχει τις διοικητικές διαδικασίες όταν ο κρατούμενος ανήκει σε εγκληματική οργάνωση ή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα, η κινδυνη από το προφίλ, το εγκληματικό των κρατούμενων που ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις μπορούν ε, να συνοσπιστούν στο εξή. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τους ε, κρατούμενους ε, αυτούς, διότι μπορεί είτε να προχωρήσουν σε διαφορά απέναντι στο προσωπικό των, των φυλακών, για παράδειγμα, είτε απέναντι στους άλλους κρατούμενους, να χρησιμοποιήσουν μεθόδους προσιλητισμού είτε να δημιουργήσουν προβλήματα για την ασφάλεια της φυλακής, είτε να έχουν επαφές με άλλες οργανώσεις εγκληματικές, το οποίο τους βοηθάει τους κρατούμενους αυτούς να ενημερώνονται για άλλες τεχνικές ή για άλλες στοιχεία που έχουν να κάνουν με το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης μπορεί να υπάρξει προσπάθεια απόδρασης από τις φυλακές εξαιτία συνεννόησης που μπορούν να έχουν με άλλα μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Ή πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι μέσα στη φυλακή έχουμε την αναπαραγωγή των ε, ίδιων μορφών εξουσίας όπως έχουμε και στην κοινωνία. Οι εγκληματικέ οργανώσεις επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι εξακολουθούν να ελέγχουν τα μέλη τους που είναι κρατούμενοι στις φυλακές. Και έτσι μπορούν και μεταφέρουν τις ίδιες δομές και μέσα στη φυλακή. Στη χώρα μου, οι κρατούμενοι χρησιμοποιούνται επίσης για να επιτευχθούν και πολιτικά ωφέλη στο εξωτερικό. Γίνεται δηλαδή εκβιασμός από τις οργανώσεις αυτές στην εξουσία. Έχουμε λοιπόν οργανωμένο έγκλημα στην χώρα μου στην Ισπανία και θα αναφερθώ σε αυτό πρώτα και μετά στην τρομοκρατία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στην Ισπανία έχει υπάρξει και υπάρχει ακόμα αυτόχθονη τρομοκρατία η οποία έχει επιβιώσει πάρα πολύ πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεν προχωράει σε τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά ε, παρόλα αυτά έχει επαφές με τους κρατούμενους. Η δραστηριότητα πάτος του σοφρονιστικού συστήματος προβλέπει κάποιες δράσεις όταν πρόκειται για τέτοιους κρατούμενους συνδεμένους με την τρομοκρατία. Και έχει δημιουργήσει μια ειδική οργανωτική δομή προκειμένου να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους εγκληματικότητα μέσα στις φυλακές. Γι' αυτό ακριβώς στη χώρα μου η σοφρονιστική ε, δίκηση εξαρτάται από το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. υπάρχουν ε, έλεγχοι μέσω πληροφορική όσον αφορά τους κρατούμενους ε, αυτούς και υπάρχει ειδική κατάρταση του προσωπικού των φυλακών προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε επίσης και ένα ειδικό φάκελο για τους κρατούμενους ειδικού ελέγχου, όπως τους λέμε. Και εκεί συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για όλους τους κρατούμενους οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές εξαιτίας ε, οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας. Η ασφάλεια του κράτους έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν έχουμε να κάνουμε με κλιματικές οργανώσεις που έχουν ε, δυνατότητες ε, ε, προσφυγής στην βία από την οποία κινδυνεύουν οι πολίτες μας. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε και ειδικό συντονισμό με όλες τις δυνάμεις ασφάλειας του κράτους που μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες και να λάβουν σοφρονιστικές αποφάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν. Έρχομαι τώρα στα προγράμματα παρέμβασης που έχουμε για τους κρατούμενους που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Προσπαθούμε να πετύχουμε τον ε, έλεγχο και την απομάκρυνση των κρατούμενων από τις οργανώσεις τους. Και αυτό ε, βάζοντας τους κρατούμενους σε διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επαφές μεταξύ τους και ώστε στα διάφορα αυτά σοφρονιστικά κέντρα να μπορέσουν να απομακρυνθούν από τις κλιματικές δραστηριότητε. Υπάρχουν επίσης έλεγχοι της επικοινωνίας και των επαφών που έχουν οι κρατούμενοι αυτοί με άλλους κρατούμενους ή εκτός φυλακής. Ελέγχεται το υλικό πληροφορικής, όπως επίσης γίνεται εντατική παρατήρησή τους προκειμένου να διαπιστώσουμε αν έχουν επαφές με επαγγελματίες, με άλλους κρατούμενους, ε, ποιος έχει ηγετικό ρόλο και τι σχέσεις επίσης έχουν με άλλους κρατούμενους από άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Συγχρόνως, περιορίζουμε και τις εξόδους. Είναι πολύ σημαντικό να ειδικευτούν οι αρμόδιοι του σοφρονιστικού συστήματος για τέτοιου είδους κρατούμενους. Γι' αυτό και υπάρχουν ειδικά προγράμματα κατάρτισης. Στην Ισπανία εξαρτώνται κάπου 60.000 κρατούμενοι από την Γενική Σοφρονιστική Δίκηση. Πρέπει όμως να σας πω επίσης ότι στη χώρα μου υπάρχει και σοφρονιστική αρμοδιότητα στην Καταλωνία, που είναι μια ισπανική περιφέρεια, που διαχειρίζεται περίπου 10.000 κρατούμενους. Πιο συγκεκριμένα, από τα στατιστικά δεδομένα, τα πιο πρόσφατα που έχουμε όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, στην Ισπανία έχουμε... διακόπτει ο πρόεδρος. Πιο αργά να μιλάτε παρακαλώ για να σας προλαβαίνει η διερμηνία, λέει πρόεδρος. Συνεχίζει ο μιλητής. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε 368 κρατούμενους του οργανωμένου εγκλήματος, από τους οποίους 357 είναι άντρες και 11 γυναίκες. Από πού προέρχονται, κυρίως από την Ισπανία 147, από την Κολομβία 80, από την Ιταλία 19, 7 από την Τουρκία, 10 από τη Βενεζουέλα, 5 από τη Ρουμανία, 5 από το Μεξικό, 3 από το Μαρόκο και οι υπόλοιποι είναι από άλλες ε, υπηκότητες, λιγότεροι βέβαια από άλλες χώρες. Οι καταδίκες ως επιτοπλίστων είναι 9 με 10 χρώματα, ε, χρόνια. Και επικεντρωνόμαστε κυρίως, μιλάμε δηλαδή για εγκλήματα που έχουν να κάνουν για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, για παράνομη μετανάστευση, για λαθρεμπόριο όπλων, για νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, για λαθρεμπόριο οχημάτων, για εμπόριο παιδιών, για διαφθορά, για αγοροπολισία παράνομου ραδιενεργού υλικού, για πορνεία, για λαθρεμπόριο έργων τέχνης, για λαθρεμπόριο υποπροστασία ζών και για κλίματα κατά της ε, ιδιοκτησίας. Πιο πρόσφατα έχουμε και απαγωγές, χωρίς όμως να είναι πολιτικού χαρακτήρα. Σε ποιες ε, περιοχές τώρα παρατηρούνται τα εγκλήματα αυτά, κυρίως στις ακτές και στις μεγάλες πόλεις. Σε σχέση τώρα με τους κρατούμενους, των ε, οποίων η εγκληματική δραστηριότητα έχει να κάνει με τον ε, αυτόχθονο, αυτόχθονη τρομοκρατία είναι 154. Ως επιτοπλίστων οι καταδίκες είναι πάνω από 20 χρόνια κάθεξη. Σε σχέση τώρα με άλλες ε, τρομοκρατικές ε, οργανώσεις διεθνού χαρακτήρα που συνδέονται με την Τζιχάτ για παράδειγμα, τα στοιχεία που έχουμε είναι του Ιουλίου και έχουμε 51 κρατούμενους. Οι καταδίκες τους είναι 9 με 20 χρόνια φυλάκιση. Από πού προέρχονται από χώρες που βρίσκονται κοντά σε εμά, Μαρόκο κυρίως, αλλά και στη συνέχεια Πακιστάν, Αλγερία, Συρία κλπ. Θα προσπαθήσω τώρα, επειδή μου έχετε δώσει λίγο χρόνο, θα προσπαθήσω τώρα να αναφερθώ στις οχρονιστικέ πρωτοβουλίες για την ασφάλεια που έχουμε υιοθετήσει για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις ε, συμβάντων, επεισοδίων στα οποία έχουν ε, πρωταγωνιστήσει οι κρατούμενοι μας. Μόνο μία τραπέτευση έχουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Η στοιχεία όσον αφορά τη χειραγώγηση, τη διαφθορά που προσπάθησαν να πετύχουν οι κρατούμενοι απέναντι στο προσωπικό των φυλακών ε, είναι ασήμαντα τα δεδομένα που έχουμε. ούτε έχουμε και αρνητικά δεδομένα, απειλές για παράδειγμα, η προσπάθεια για ε, διαφθορά, οι απειλές απέναντι σε μάρτυρες. Στις περιπτώσεις αυτές έτσι κι αλλιώς δεν ε, πέτυχε τίποτα απέναντι στο σοφρονιστικό σύστημα. Παρόλο που όπως γνωρίζετε η ομάδα αυτή κρατούμενων συνήθως έχει χρήματα και μπορεί να πληρώσει και πολύ καλούς ε, δικηγόρους. Οι προσπάθειές μας προσανατολίζονται στην επανένταξη. Δυστυχώς όμως εκεί δεν έχουμε πετύχει πολύ. Και αυτό γιατί συνήθως οι εγκληματικές οργανώσεις βρίσκουν άλλες μεθόδους και έτσι τελικά οι κρατούμενοι οι οποίοι έμειναν στη φυλακή για λίγα χρόνια ή για τους οποίους υπήρχε στέρηση ελευθερίας ε, χωρίς ε, όμως να βρίσκονται στη φυλακή, αυτοί αναμειγνύονται και πάλι στο οργανωμένο έγκλημα. Και έχουμε βέβαια και τη θεωρία γενικότερα των υποτροπιαζόντων. Εμείς θέλουμε μια σοφρονιστική πολιτική η οποία να βοηθάει τους κρατούμενους ε, αυτούς. Και γι' αυτό και έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα με το οποίο προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την, ε, τον έρθει σε πέρα, να φέρει σε πέρα στην ποινή του ο κρατούμενος και τους ε, προσφέρουμε κατά τη διάρκεια της κράτησής τους φορά προγράμματα απασχόλησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην περίπτωση της τρομοκρατίας, τα χαρακτηριστικά των κρατούμενων, το κατά πόσο αναγνωρίζουν τη βλάβη που έχουν προκαλέσει, κατά πόσο έχουν αποποιηθεί τις ε, πεπιθήσεις τους. Αυτά αποτελούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των κρατούμενων, βάσει των οποίων ακολουθούμε και συγκεκριμένη στρατηγική. Στην περίπτωση της οργάνωσης μάλιστα η οποία έχει στερήσει τη ζωή από πάρα πολλούς Ισπανούς, η οργάνωση αυτή παραμένει, ενισχύει και έχει και κάποια κοινωνική στήριξη και γι' αυτό οι κρατούμενοι από την οργάνωση αυτή παραμένουν στη συγκεκριμένη δομή. Εμείς πάντως έχουμε αυτό το πρόγραμμα παρέμβασης με θετικές δράσεις. Προσπαθούμε να απομακρύνουμε τους κρατούμενους από τις οργανώσεις τους και από την επιρροή των οργανώσεών τους. Βέβαια, μέσα σε πλήρη νομιμότητα προσπαθούμε να προσφέρουμε στους κρατούμενους αυτούς ένα κατάλογο δραστηριοτήτων οι οποίες τους διευκολύνουν να απομακρυνθούν από την τρομοκρατική τους οργάνωση. Ζητώ συγγνώμη από τους μεταφραστές, λέει ο μιλητής, γιατί προχώρησα τόσο γρήγορα. Αλλά προσπάθησα να τηρήσω το χρόνο μου, βλέπετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την υπομονή σας και για τον ενδιαφέρον που δείξατε στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δώσουμε τώρα το λόγο στον Τζόνας Γκρίντεν, από ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εσείς έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή και μετά θα ανοίξουμε τον γύρο των ερωτήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να ε, ασχοληθώ να μιλήσω για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Ε, ε, ο κύριος Αλφάνο ε, και η Επιτροπή μας κάλεσαν και χαιρόμαστε πάρα πολύ, όπως επίσης και για την επιστολή του κυρίου Σούλτς που αναφέρθηκε και αυτό στο ίδιο. Τρία θέματα θέλω να τυλίξω να γνωρίζετε καταρχήν τι είναι η δική μας, ε, τι είναι ο οργανισμός μας, τι έχουμε κάνει για το οργανωμένο έγκλημα και βέβαια μετά θα ήθελα να παρουσιάσω διάφορα στοιχεία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Καταρχήν, τι είναι η ε, δική μας, τι είναι ο οργανισμός μας. Στη Βιέννη είμαστε, βρισκόμαστε, έχουμε λοιπόν ε, το καθήκον να εφαρμόζουμε το κοινοτικό δίκαιο και οποτεδήποτε γίνεται αυτό να είναι συμβατό με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεύτερον, λειτουργούμε προληπτικά αν μπορώ να το πω αυτό. Έχουμε αυτή την εντολή να λειτουργούμε προληπτικά για να συντάσσουμε συγκριτικές μελέτες που βασίζονται σε κοινωνικο-οικονομικές μελέτες. Ε, ε, έχουμε το πενταετές πρόγραμμα το οποίο συνέταξε η Επιτροπή και συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και έχουμε επίσης και την εντολή αντίδρασης να τοποθετηθούμε οποτεδήποτε καλούμεθα να το πράξουμε αυτό από οποιονδήποτε οργανισμό, προφανώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να αντιδρούμε για ε, σχέδια νομικών πράξεων, αλλά και άλλων θεμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πενταετές ε, ε, πρόγραμμα, στην πενταετή εντολή. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη βάση και επειδή υπάρχουν αυτά, γι' αυτό ήρθαμε και εμείς εδώ σήμερα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ο Οργανισμός των Πολιτών Δικαιωμάτων, ο δικός μας οργανισμός, τι ακριβώς έχει κάνει σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Αν θέλετε, ε, τίποτα το συγκεκριμένο ως τέτοιο, αλλά και πάρα πολλά που έχουν άμεση σχέση με ε, θέματα. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Συγκριτικές μελέτες και εγχειρίδια Έχουμε δημοσιεύσει μια έκθεση για την εμπορία παιδιών. Έχουμε ένα εγχειρίδιο για τα προφίλ, ε, για ε, τις προκαταλήψεις που υπάρχουν σχετικά με τα εθνικά προφίλ που χρησιμοποιεί η αστυνομία, πότε είναι καλό και πότε είναι αρνητικό. Κατόπιν έχουμε μελέτη για τις διακρίσεις. Ε, τώρα τρέχει μια μελέτη για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων. Το ψάχνουμε αυτό στις 27 χώρες πλάς συν μια η Κροατία. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τι λειτουργεί καλά, έχοντας κατά νου να καθοριστούν στρατηγικές ε, που είναι αποτελεσματικές και τι μπορεί να βοηθήσει τα θύματα. Και βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει είναι η αντιμετώπιση των θυμάτων της βίας. Ε, αυτό είναι κάτι που κι εσείς από τη Μέση διάταξη το έχετε εξετάσει. Επίσης έχουμε ασχοληθεί με την ε, παράνομη εισδοχή μεταναστών. Υπάρχουν ε, κάποια προγράμματα που αφορούν ε, σε υπηκόους τρίτων χωρών, δικαιώματα μεταναστών, παράνομων κυρίως μεταναστών. Προτιθέμετα του χρόνου να ασχοληθούμε με σοβαρές μορφές εκμετάλλευσης της εργασίας. Τότε ψάχνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Εργασίας. Τώρα, πάμε λίγο στις ε, αντιδράσεις. Πότε τοποθετηθούμεθα ε, όποτε μας το ζητούν. Για το PNR μας το ζήτησαν. Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πολύ καλά το θέμα. Και υπάρχει δική μας γνωμοδότηση, δημοσιεύτηκε και πέρυσι, ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή εντολή ανάκρισης. Ένα άλλο στοιχείο ε, δραστηριοτήτων μας έχει σχέση με την ανταλλαγή και τη συνεργασία. Ε, ορισμένοι οργανισμοί με τους οποίους ε, συνεργαζόμετα είναι αυτή που θα έχετε ακούσει τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε τη Frontex, ε, συνεργαζόμαστε μαζί τους ε, για την εκπαίδευση παραμεθόριων φυλάκων, να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματά τους, να υπάρχει στρατηγική θεμελιωτών δικαιωμάτων. Ε, συνεργαζόμεθα με την ΣΥΠΟΛ και εκεί έχουμε ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης το οποίο χρησιμοποιείται σε αστυνομικές ε, ακαδημίες. Ε, με τη Europol συνεργαζόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα και υπάρχουν εδώ δύο συνάδελφοι ε, στην ε, Χάγη έχουμε στις πολλά θέματα που μας αφορούν ε, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση εργασίας και προστασία δεδομένων είναι μια ανταλλαγή απόψεων σε τακτική χρονική βάση και επίσης συμμετέχουμε και στη συνεργασία δικαστικών αρχών και εσωτερικών υποθέσεων τελευταίο θέμα για το τι ακριβώς κάναμε έχει σχέση με το πάγωμα ε, κεφαλαίων, ε, δίμευση ε, παράνομων κερδών. Συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν για τα θέματα αυτά και θα συνεχίσουμε. Πάω τώρα στο τρίτο σημείο της παρέμβασής μου και αυτή είναι και η ουσία της. Θεμελιώδη δικαιώματα και οργανωμένο έγκλημα. Όπως είπα στην αρχή θα είμαι πάρα πολύ σύντομος επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Η σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων προβλήθηκε από προλαλήσαντες ε, και είναι σημαντική, ε, σημαντική βέβαια η πρόληψη για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα και γενικότερα το έγκλημα και έχει σχέση με τα δικαιώματα αυτών που πλήττονται από τέτοιου είδους εγκλήματα αλλά ε, εδώ πρόκειται και για τα δικαιώματα των υπόπτων, ε, των καταδικαστέντων και των μαρτύρων. Εδώ γίνεται λόγος για μια ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της. Επίσης ε, γίνεται λόγος για την Ευρώπη της δικαιοσύνης και της ελευθερίας ε, και προβάλλονται προφανώς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίζει ε, τα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη ξεχωριστά το καθένα από αυτά και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που θέλουμε να προβάλλουμε. Αν δούμε λιγάκι την ομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου και αυτή του Λουξεμβούργου που είναι τα δύο πιο σημαντικά δικαστήρια, αν δούμε λιγάκι την ομολογία τους, ε, θα ήθελα να προβάλλω οκτώ τομείς ε, όπου εξέτασαν περιπτώσεις με σαφή αναφορά στο οργανωμένο έγκλημα. Δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα, ε, λογοκρισία επιστολών φυλακισμένων, προστασία δεδομένων, συνθήκες ε, κράτασης, ε, απομόνωση, πάγωμα και δίμευση περιουσιακών στοιχείων, δίκαιη δίκη αλλά και άλλα στοιχεία όπως δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, δικαιώματα των θυμάτων των εγκλημάτων, παρακολούθηση, τηλεφωνική παρακολούθηση, εκχώρηση εξαιρέσεις, ε, πότε μπορούν να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ε, σε σοβαρές περιπτώσεις, αντιτρομοκρατία. Είδαμε τα δικαιώματα της, ε, των κατηγορουμένων και ανακεφαλαιώνοντας, νομίζω, αν θέλετε, μπορώ βέβαια να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά έχοντας κατά νου την ώρα και τις άλλες υποχρώσεις, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω και να αναφερθώ λιγάκι σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ πρόκειται για την αναλογική χρήση της εξουσίας σε αναλογία με τον επιδιωκόμενο στόχο. Δεν είναι ένα τυχαίο σύστημα δικαιωμάτων, ας πούμε, των υπόπτων, αλλά πρόκειται για την ε, εξισορρόπηση στόχου και εξουσίας. Αναφέρθηκα λοιπόν στην ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και αυτή του ε, Λουξεμβούργου για να δείξω ότι ε, είναι πολύ σημαντικές οι αποφάσεις τους. Ε, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εμείς καταφεύγουμε και σε άλλες ομολογίες Οποτεδήποτε καλούμε θα να αναλύσουμε νομικές καταστάσεις. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βασανιστήρια, το ξέπλυμα του χρήματος. Υπάρχει η Επιτροπή των Ηνωμένων κατά των βασανιστήριων και πέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι οργανισμοί, υποοργανισμοί των ΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας και αυτός ε, έχει τις δικές του ερμηνείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς, οποτεδήποτε χρειάζεται, επικαλούμεθα αυτά τα έγγραφα. Τελειώνοντας λοιπόν, Θέλω να πω το εξή. Ε, εξέτασα τρία θέματα. Το τι έχουμε κάνει με αυτό, τι είναι ο οργανισμό βέβαια και πώς ε, γίνεται η διασύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι καθοριστικό σημείο και στοιχείο στον τρόπο αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Ο οργανισμός μας ε, μπορεί να βοηθήσει ε, όπως σήμερα και σε άλλες συναντήσεις μετά από αίτημα εμείς ε, δεν έχουμε προληπτική εντολή, ε, πρέπει να κληθούμε να ε, σχολιάσουμε για ε, νομοθεσίες, νομολογίες ή άλλα έγγραφα. Ε, όπως σας είπα, επικαλούμε τα νομολογία αλλά και εμπειρογνωμοσύνη ειδικών φορέων. και καταλήγουμε, πιστεύω, σε ισορροπημένες αναλύσεις. Εγώ σήμερα απλούστευσα λιγάκι τα θέματα της νομολογίας. Σας ανέφερα απλά που τα θεμελιώδη δικαιώματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Και αυτό είναι και δουλειά της Επιτροπής σας. Το τελευταίο, τρίτο και τελευταίο στοιχείο που θέλω να πω είναι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που λαμβάνετε υπόψη σας τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, και τα, ε, τα προβάλλετε στο τόσο σημαντικό έργο που επιτελείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκριμχέντεν και τον κύριο Καστιγέχο. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας, γιατί οι απόψεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη συνέχιση και των δικών μας εργασιών, για την κατάρτιση της τελικής έκθεσης του κυρίου Γιακολίνου. Και σε αυτό το κλάστερ θέλαμε να προσεγγίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα γιατί Εμεί ε, θέλουμε να σεβαστούμε πλήρω τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θέλουμε και να κατανοήσουμε πώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ευνομικαστικά καταστήματα με σκοπό την παιδεία δηλαδή και να λάβουμε υπόψη τα θύματα που έχουν αδικηθεί αλλά και ότι μπορεί να εκτιθεί τελικά η ποινή και να υπάρχει στη συνέχεια επανένταξη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα της ε, επανεκπαίδευσης ως στόχο της κάθεξης. Μπορείτε να πάρετε το λόγο για να κάνετε τις ερωτήσεις, ε, για να έχουμε και περισσότερο χρόνο για τις απαντήσεις. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιακολίνο καταρχήν. Είναι και ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα μόνο εν μέρη την πρώτη παρέμβαση του κυρίου Καστιγέχο, που είναι επικεφαλή ε, τη ε, διοίκηση των σοφρονιστικών καταστημάτων, ε, όμως άκουσα ολόκληρη την παρέμβαση του άλλου μιλητή, ο οποίο προέρχεται από τον οργανισμό μελλοντών δικαιωμάτων. Να περάσω στην ερώτηση. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να παντρέψουμε ε, το σεβασμό των ε, δικαιωμάτων ε, κάποιου που πρέπει να εκτίσει μια ποινή, κυρίω όταν η ποινή αυτή πρέπει να εκτιθεί σε μια φυλακή όπου υπάρχει υπερπληθυσμό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Θέλουμε μια δίκαιη δίκη και φυσικά απαιτείται και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κύριε Διευθυντά, στην παρέμβασή σας δεν αναφερθήκατε στο σκληρό καθεστώς, το καθεστώς της απομόνωσης ε, αν θέλετε, έχουμε κάποιες άλλες πραγματικότητες, ε, προέρχονται ε, από άλλες χώρες. Ε, θέλουμε να δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το καθεστώς της απομόνωσης δηλαδή να τίθενται σε απομόνωση οι μαφιόζοι για να μην μπορούν να συνεχίσουν ε, το ρόλο τους μέσα στη φυλακή. Τι σκέφτεστε για το καθεστώς αυτός και να στραφώ και στον κύριο Κρυμχέντεν να μας πείτε αν ε, θέλουμε ένα περιορισμό, μια περιστολή ο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις όπου ε, θα διασφαλίσουμε καλύτερα με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Νιτοντάν για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν και δύο παρουσίασει εξαιρετικές και ιδιαίτερα πολύτιμέ για μα. Ε, σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε τόσο μακριά για να φτάσατε μέχρι εδώ. Θα ξεκινήσω με τον Ισπανό μιλητή. Έχω πολλές ερωτήσεις. Ποιο ποσοστό σε έγκλειστον ε, τελικά πάνε στο πανεπιστήμιο και μαθαίνουν και πανεκπαιδεύονται. Δηλαδή, τι ελπίδα έχουμε για αυτή την επανεκπαίδευση και πόσους μπορούμε να επανεκπαιδεύσουμε έτσι ώστε να περιορίσουμε αυτό το τόσο επικίνδυνο πρόβλημα. Και δεύτερον, αυτό που θέλει να ξέρει αυτή η Επιτροπή είναι πώς μπορεί να καταπολεμήσει τους ανθρώπους αυτούς καλύτερα. Αυτό θα είναι το συμπέρασμα του χρόνου, όταν θα συντάξουμε την εκθεσή μας, εσείς, δηλαδή στο δικό σας τομέα. Τι θα θέλετε να δείτε, τι μπορεί να κάνει καλύτερη η Ευρώπη. Και αν μου πείτε, κοιτάξτε, εγώ, ε, αν μας πείτε τώρα, ε, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί εγώ απλώς είμαι διοικητής των φυλακών, όμως μπορείτε να βγείτε από αυτό το ρόλο και να μας πείτε τι θα μας συστήνατε, τι θα ήταν χρήσιμο ε, κατά τη δική σα άποψη θα μα βοηθούσε πάρα πολύ. Στο ό,τι αφορά τώρα στον εμπειρογνωμένο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, είναι πολύ σημαντικό ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον πολιτισμό μα και για την κοινωνία μα και σα ευχαριστώ για εσά είπατε. Αλλά θα σα θέσω την ίδια ερώτηση, τι θα πρέπει να συστήσουμε του χρόνου, ποιε αλλαγέ, Τώρα, αν, πιστεψ... αν μας πείτε κι εσείς, α, δεν θα τοποθετηθώ εγώ γιατί εργάζομαι σε εργαζόμενο και εσείς βγείτε από αυτό το ρόλο και να μας δώσετε τη συμβουλή σας ως πολίτης με εμπειρία. Τι θα πρέπει να συστήσει η Επιτροπή μας, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που άκουσα από ένα αστυνομικό νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα που εργάζεται στο διαδίκτυο. Είναι παράνομο στην Ευρώπη, μου είπε, να ε, προσπαθήσουμε να παγιδεύσουμε στο διαδίκτυο του εγκληματίες. Αν ε, δυσδύσει κάποιος σε μια συμμορία μέσω διαδικτύου ε, και αν ε, τους ε, παρακολουθεί από εκεί και τους βάλει κάποιο δόλωμα, τότε η αστυνομία παρανομεί, γιατί δεν σέβεται την ιδιωτικότητά του ενώ στην Αμερική είναι αυτό απολύτως νόμιμο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα και νομίζω ότι εδώ είναι σαν να φερούμε κάποια εργαλεία από τον εαυτό μας, ε, σαν να καθιστούμε τους αυτούς μας ανάπηρους. Έτσι λοιπόν, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συστάσεις, αν βγείτε από το ρόλο σας και μπορείτε να μας δώσετε τέτοιες συστάσεις, θα είναι πολύ χρήσιμο για μας. Ευχαριστώ κύριε Νιουτοντάν για το ΕΛΚ. Η κυρία Ματιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο μιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, ομιλίες τους. Κύριε Καστιγιάγο, Το Ισπανικό Σοφρονιστικό Σύστημα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Στη Γαλλία έχουμε κάποιες δυστυχείς υποθέσεις. Πριν 15 χρόνια, παραδείγματο χάρη, ε, οργάνωνε ένας κρατούμενος διακίνηση κοκαίνης και όταν ε, βγήκε από τη φυλακή ε, είχε ένα πολύ οργανωμένο λαθρεμπόριο και το θυμόμαστε ακόμα και επίσης, εγώ έχω επισκεφθεί κάποια σοφρανιστικά καταστήματα στη Γαλλία και είχαμε τη δυσάρεστη έκπληξη να δούμε στο διαδίκτυο, μάλλον, μάλλον με τη βοήθεια κάποιου κινητού, είχε περάσει ίσως κάποια κάρτα μέσω κάποιου επισκέπτη ή φαντάζομαι ότι αφήθηκε να διαφθαρεί κάποιος δεσμοφύλακας. Ε, είχαμε λοιπόν δει ένα τρομερό μήνυμα κάποιου κρατούμενου προς την οικογένεια του θύματος. Και ελπίζω στην Ισπανία να μην βλέπετε τέτοια γεγονότα, όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Ελπίζω να τα καταφέρνετε, αλλά πώς καταφέρνετε να έχετε κάποιους δεσμοφύλακες αλλά και δικηγόρους που να μην είναι διεφθαρμένοι. Που ε, έχουν πραγματικά τη δέουσα συμπεριφορά, την σέβονται τη δεντολογία. Κοιτάξτε, σε εμά ε, στη Γαλλία μερικές φορές βλέπουμε να υπάρχουν ε, διεφθαρμένοι αξιωματούχοι. Και μας είπατε ότι υπάρχουν και κάποιες γυναίκες ε, που είναι έγκλειστες ε, για οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε την ισότητα παντού, αλλά βλέπουμε ότι ε, οι γυναίκες δεν είναι και τόσο παρούσες και τόσο το καλύτερο. Γιατί όμως, αναρωτιέμαι, γιατί έχουμε σχεδόν μόνο άντρες οι οποίοι συλλαμβάνονται για οργανωμένο έγκλημα. Αυτή είναι η ερώτησή μου και για τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Συνεχίστε, έχετε πάρα πολλή δουλειά στον τομέα σας. Και εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στην Κομισιόν Ελέγχου των Προπολογισμών. Βλέπουμε πόση δουλειά κάνετε. Καλό κουράγιο λοιπόν και υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καστιγιάχο για την παρουσίασή του, καθώς και τον κύριο Κλίντεχεντεν. Κύριε Καστιγιάχο, να σας ρωτήσω. Αναφερθήκατε εσείς ε, πιο συγκεκριμένα για τη μάθηση, για την εκπαίδευση. Είναι μια μακρά εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα έτη. Τώρα όμως περνάμε σε ένα νέο στάδιο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αυτές τις νέες προτάσεις που θέλουμε να προωθήσουμε. Όμως, τι θέλω εγώ να σας ρωτήσω. Καταρχήν, η Ισπανία, και αυτό μας ανησυχεί και εδώ, ήδη φαίνεται ως ένα τόπος ε, όπου αναπαύεται η μαφία. Δηλαδή εδώ και πολύ καιρό έχει σχολιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι τα πιο σημαντικά κτυπήματα και από βίε μαφιόζικες ομάδε είναι στο εξωτερικό αλλά πηγαίνουν ε, μετά ε, στην Ισπανία, στις ισπανικές ε, ακτές για να ε, αναπαυτούν, ε, αν λέτε. Όμως, ε, λοιπόν, θα ήθελα να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό και σε ό,τι αφορά αυτό το boom στις κατασκευές που έγινε, αυτή την άνθηση ήταν ένα μέσο για να κυκλοφορήσει το βρώμικο χρήμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω βάσει της εμπειρίας σας είστε και υπεύθυνο και ε, των σοφρονιστικών καταστημάτων, αλλά έχετε και ευρύτερη εμπειρία στον τομέα ε, του Υπουργείου Συντερικών. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Τώρα, να σας ε, ρωτήσω στην κατάσταση που βρισκόμαστε, τι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των φυλακών. Βλέπουμε όμως ε, ότι η δικαιοσύνη δεν εφαρμόζεται όπως ε, πρέπει. Βέβαια νομίζω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση τελευταία και για τους σπόρους που έχουμε για τα σοφρονιστικά καταστήματα συγκριτικά. Ξέρετε τι υπάρχει και στο εξωτερικό. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία Ε, για να αντιμετωπίσουν οι φυλακές ε, αυτούς τους βίαιους ανθρώπους. Και σε ό,τι αφορά τώρα τη σχέση μεταξύ όσων εργάζονται στις φυλακές ε, και των αγγλίστων για αυτούς τους επικίνδυνους έγκλειστους, έχουμε και τα μέλη της Τζιχάντ, Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια γενική σύσταση σε σχέση με την εκπαίδευσή τους, με την κατάρτισή τους και να δώσουμε καλύτερα μέσα ε, στους εργαζόμενους στις φυλακές, στα σοφρονιστικά καταστήματα. Τι πιστεύετε εσείς. Μάλιστα, διέστε μέρα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ εκτίμησα τις παρουσιάσεις των δύο προσκεκλημένων μας. Του συγχαίρω και θα κρατήσω τα όσα είπαν για το προσωπικό μου αρχείο. Σε κάποιο άλλο στάδιο, φάση της ζωής μου, είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η αναπαραγωγή των δομών εξουσίας της κοινωνίας μέσα στις φυλακές. Πώς το καταπολεμάτε αυτό. Πώς καταπολεμάτε δηλαδή την αναπαραγωγή αυτή των δομών εξουσίας. Παράδειγμα. Εσκοβάρ. Κολομβία. Καρτέλ. ο Μεξικό. είστε Βάγια Δεκάουκα. Όταν αυτοί μπαίνουν στη φυλακή, εξακολουθούν να οργανώνονται. Εξακολουθούν να παραβιάζουν τον νόμο και να αναπαραγάγουν τις ίδιες δομές. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ανεξάρτητα τώρα από τα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή του το σοφρονιστικό σύστημα, θα ήθελα να μας πούτε λιγάκι τι μπορεί να γίνει ή τι κάνετε για να αποφευθεί αυτή η αναπαραγωγή των ίδιων δομών μέσα στη φυλακή. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπορσελίνο, δύο λεπτά. Κοιτάξτε την ερώτηση που ε, θέλω να βάλω, την, να υποβάλω, την έχει υποβάλει ο κύριος Γιακολίνο. Αλλά ε, ο συνάδελφος που μόλις μίλησε με βοήθησε στο να κάνω και εγώ την ερώτησή μου. Έχουμε το άρθρο 141α ε, στην ε, Ιταλία κάθριξη προβλέπεται για διάφορες ε, μορφές ε, εγκλημάτων. Αυτό το άρθρο, το 141α, επικρίνεται πολύ συχνά ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απορρέει όμως ακριβώς ε, από αυτό που είπε η συνάδελφος, δηλαδή Θέλουμε να αποφύγουμε μέσα στη φυλακή να αναπαράγονται οι ίδιες ισορροπίες εξουσίας που υπήρχαν εκτός φυλακής. Εσείς για αυτό το 141α ε, τι ακριβώς πιστεύετε που πρόκειται για περιορισμό ατομικών ελευθεριών. Δεν πιστεύετε κι εσείς ε, ότι αυτή η διάταξη εφόσον μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που θα ωφελούσε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Σμιτ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τις δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Προς τον κύριο Γκρίμιν ε, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι τελειώσαμε και οι δύο το ίδιο πανεπιστήμιο ε, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, University of London. Αυτό κάτι σημαίνει, είναι υπεραξία. Η ερώτησή μου είναι η γενικής φύσεως. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σωστή όπως έχει συνταχθεί. Αναφερθήκατε στο PNR. Εμείς εδώ έχουμε ασχοληθεί για πολύ καιρό με το PNR και ε, δίστανται οι απόψεις επ' αυτού. Επίσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση για το SWIFT, για τη μεταφορά τραπεζικών δεδομένων στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Και σύμφωνα με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αυτά ε, τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιήθηκαν για να διαλευκανθούν ε, υποθέσεις. Για τους πιο αγαθούς αξίζουν όλα αυτά. Και πιο γενικά να το πω. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την ομοθεσία στην Ευρώπη είναι ανάλογος ε, προς το φαινόμενο. Κυρία Χιμένες, θέλω να ευχαριστήσω τους ε, δύο μιλητές για την παρουσία τους εδώ και θα ήθελα να σας πω ότι εκτιμώ και τα όσα είπατε και οι δύο και που μιλήσατε για τα θύματα των εγκλημάτων. Από τότε που έφτασα σε αυτό το κοινοβουλίο, Πραγματικά το θέμα των θυμάτων ήταν από τα πλέον ξεχασμένα και πριν λίγες, σέρες, ε, ε, μέρες εγκρίναμε την οδηγία για την υποστήριξη των θυμάτων. Είμαι συγγήτρια εγώ για την οδηγία αυτή και νομίζω ότι πετύχαμε σημαντικά ε, δικαιώματα όπως το χάρη να προσφέρουμε υποστήριξη στα θύματα, μετάφραση, να εγκριθεί ένα κέντρο υποστήριξης για τα θύματα. Αλλά θέλω να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Κρυμχεντέν. Αν πιστεύετε ότι τα όσα κάνουμε, αν αυτή η οδηγία μπορεί να συμβάλλει στο να πιστέψουν οι πολίτες ότι υπάρχει μια κοινή δικαιοσύνη και ένας κοινό χώρος ασφάλειας και προστασίας, γιατί εγώ νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και για ε, να συνδέσω και μία ερώτηση με την άλλη. Θα ήθελα να σας πω εσείς πιστεύετε ότι τα θύματα όλο ένα και περισσότερο αρχίζουν να μην ε, εμπιστεύονται ότι υπάρχει κάθριξη της ποινή, δεν έχουν εμπιστοσύνη. Παραδείγματο χάρη, ε, έχουμε τη θανατική ποινή. Εγώ είμαι κατά τη θανατική ποινή. Πάντα ε, ήμουν ενεργή και στην Ιαπωνία για να καταπολεμήσουμε τη θανατική ποινή. Και επίση είμαι κατά και τη ισόβια κάθριξη όμως ε, όλα αυτά ε, μάλλον πρέπει το θύμα να πιστεύει ότι θα εκτιθεί ποινή. Αν αρχίζει το θύμα να πιστεύει ότι δεν θα εκτιθεί η ποινή ή τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει συνέπεια. Έτσι λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε ε, μια απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου κατά μιας ε, ε, Ισπανίδας ε, η οποία καταδικάστηκε σε δύο ή τρεις χιλιάδες χρόνια για τρομοκρατικές πράξεις. Όμως νομίζω ότι πέθαναν κάποιοι πάρα πολλοί νέοι, 22-23 χρονών και τώρα λένε ότι πρέπει να την θέσουν στη φυλακή και ε, τις ε, έχουν επιδικάσει να πληρώσει πάνω από 6.000 ευρώ στα θύματα. Όμως ε, πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο υποσκάπτει την αξιοπρέπεια των θυμάτων και ε, την εμπιστοσύνη που έχουν τα θύματα στη δικαιοσύνη και αν αρχίσουν τα θύματα να μην εμπιστευτούν τη δικαιοσύνη, τότε αρχίζουν τα θύματα να ζητούν θανατική ποινή και τέτοια πράγματα, γιατί δεν πιστεύουν ότι όσους έκανε κακό θα πληρώσει εδώ ε, έχουμε κάποιου που εκπροσωπούν το σαφρονιστικό σύστημα αλλά και το σεβασμό των δικαιώντων. Εσεί ε, πώ πιστεύετε ότι μπορούν τα θύματα να πιστέψουν ότι θα εκτιθεί αυτή η ποινή από του καταδικασμένου. Μάλιστα, αυτό που συνέβησαν ε, είναι τρομερά έτσι λοιπόν, ε, γιατί εδώ ε, πάλι μπορεί να υπάρχει αλλαγή των ρόλων, να γίνει το θύμα θήτης και το αντίθετο. Έτσι λοιπόν, εγώ συμφωνώ αν πρέπει να αγγιθούμε την δίκαιη αναγνώριση στα θύματα, αλλά και πρέπει να τους βοηθήσουμε να ψεύσουν στη δικαιοσύνη. Υπάρχει και, πρέπει να υπάρχει και βεβαιότητα της ποινή στην Ιταλία. Υπάρχει η εξή σκέψη Δηλαδή ότι ε, τελικά πάντα ε, την ποινή την εκτείνουν τα θύματα γιατί είναι μια ποινή η οποία διαρκεί όλη τη ζωή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καστιλέχο. Καστιλέχο, η Ισπανία θεωρείται μια από αυτές τις χώρες όπου είναι εντελώς, ε, έχει εντελώς εξαλειφθεί η μαφία και η Ισπανία είναι μία από τις χώρες όπου έχουν συλληφθεί οι περισσότεροι μαφιόζοι. Τώρα, ε, προέκυψε από τις Ιταλικές Διοκτικές Αρχές ότι οι Ιταλοί ε, μαφιόζοι που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Ισπανία έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν ε, το παράνομο έργο τους και να διατηρούν ε, την ηγετική τους θέση και από αυτές τις υποκλοπές είπαν ότι αυτοί προτιμούν να εκτείνουν την ποινή τους στην Ισπανία γιατί θεωρούν ορισμένες φυλακέ, ορισμένες σοφρονιστικά καταστήματα σαν μεγάλα ξενοδοχεία. Και το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι, που θέλω να κάνω είναι για το Σάντο Μεσάνο, τον Πόσο από την Καλαβρία, που έχει συλληφθεί πάρα πολλέ φορές στην Ισπανία. Και αυτός είχε πολύ μεγάλες ικανότητες ε, γιατί μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών. Πάρα πολλές φορές ε, έχει συλληφθεί και έχει κρατηθεί στη φυλακή Βαλντεμόρο στη Μαδρίτη από το 2000, ε, μάλλον από το στο 2004. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια αυτών των υποκλοπών εμφανίστηκε ότι μιλούσε με κάποιους από τη συμμορία του και έλεγε ότι είναι μεγάλο ξενοδοχείο η φυλακή και μπορούσε να συνεχίσει να κάνει επιχειρήσεις. Και έτσι ήταν. Ήταν πραγματικότητα αυτό, γιατί αυτό στην περίοδο της κράτησή του μάλιστα διέταξε και δολοφονίες, ε, οργάνωσε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και ε, κάθε μήνα έρχονταν στη φυλακή υπηκοοί του που συνεχίζονταν, ε, συνέχισαν να τον επισκέπτονται και να οργανώνουν ε, όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητε. Θέλω να σας ρωτήσω, έχουν ε, ληφθεί κάποιες κάποια μέτρα ασφαλεία τα τελευταία χρόνια για να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Και με τον κύριο δεν θέλω να σα ρωτήσω ποια αντίληψη έχετε εσεί για το 41α. Συχνά το 41α το βάζουμε δίπλα με το καθεστώ απομόνωση. Και πολλέ φορέ εμεί, μιλώντα με του συναδέλφου, έπρεπε να εξηγήσουμε ότι δεν είναι βασανιστήριο, αλλά και επιστήνω μια πρόσκληση εγώ εδώ, μια έκκληση. Εγώ έχω επισκεφτεί πάρα πολλέ φυλακέ και τη 01 Α, το επισκέφτηκα ε, την περασμένη εβδομάδα εκεί έχουμε πάρα πολλούς ε, επικεφαλεί της Καμόρα, της Δράγκεντα κτλ. Και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου και σε κανονικό καθεστώς και σε καθεστώς 41α εγώ είδα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου δεν γίνονται σεβαστά ε, στο κανονικό καθεστώς γιατί έχουμε οκτώ κρατουμένου σε ένα πάρα πολύ μικρό κελί και για τα άτομα αυτά είναι αδύνατο ε, να είναι όλοι μαζί όρθιοι στο ίδιο κελί, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Πολύ συχνά έχουν ε, τη δυνατότητα να κάνουν ντους μόνο τρει τέσσερι ημέρε και πρόκειται για πάρα πολύ μικρά κελιά. Όποιος όμως ε, κρατείται στο 41α, γιατί υπάρχει αναγκαιότητα τα άτομα αυτά να μην κάνουν τα ίδια που έκανε ο Μετζανό από τη φυλακή του Βαλτεμόρο, βρίσκονται ένα κελί μόνοι τους, έχουν συγκεκριμένες ειδικέ υπηρεσίες προκειμένου να αποφευχθεί τα άτομα αυτά να συνεχίζουν ε, να είναι σε διάλογο με όσους είναι εκτός της φυλακής και να μπορούν ε, να ε, λειτουργούν ως αρχηγοί της μαφίας. Ποια είναι η δική σας αντίληψη σχετικά με το κανονικό καθεστώς όπου υπάρχει πλήρης παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, του καθεστώτος απομόνωσης του 41α που θεωρείται ως ένα σκληρό καθεστώς ε, και περιορίζει την επικοινωνία με όσους είναι εκτός αφενός, αλλά από την άλλη υπάρχει απόλυτο σεβασμός των θεμελιώδων δικαιωμάτων, ε, γιατί αν βάλουμε δίπλα-δίπλα αυτές δύο πραγματικότητες, κατανοούμε πώς τα άτομα αυτά ε, ουσιαστικά βρίσκονται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τους άλλους που βρίσκονται στο κανονικό καθεστώς. Καταρχήν κύριε Καστιγέχο και κατόπιν ο κύριος Γκριμπιέντεν. Πέντε λεπτά ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Γιακολίνο ρώτησε πώς συνδυάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ε, ποινή κάθερξης. Όντως, στις ε, ισπανικές φυλακές μερικές φορές υπάρχει αίσθηση ότι πρόκειται για ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Άλλοι όμως, άλλες οργανώσεις, κυρίως τρομοκρατικές, λένε ότι οι κρατούμενοι ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Αντικειμενικά λοιπόν είναι περίπλοκο. Η ζωή στη φυλακή σίγουρα είναι σκληρή. Η στέρηση ελευθερίας είναι σκληρή. Ορισμένα άτομα τα οποία έχουν ε, προκαλέσει βλάβη στην κοινωνία βρίσκονται στη φυλακή βάσει δημοκρατικών διαδικασιών. Το μόνο που μπορώ να σας πω γι' αυτό είναι ότι εμείς τηρούμε τον νόμο. Ο κύριος Νιούτον Ντάουν τώρα είπε τι ποσοστό κρατούμενων τελικά εντάσσονται και πάλι στην κοινωνία. Εξαρτάται. Και εξαρτάται και από την ηλικία οι έγκλειστοι που βγαίνουν από τη φυλακή πιο αργά δεν ε, επαναλαμβάνουν, δεν, ε, δεν υποτροπιάζουν όσο οι νέοι. Οι τρομοκράτες βέβαια μπορεί μεν να μην υποτροπιάζουν, δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρησιμοποιούνται από την εγκληματική τους οργάνωση για, με καθαρά πρακτικούς τρόπους, γιατί τελικά δεν ε, μετανοούν ούτε καταδικάζουν τα εγκλήματά τους. Τώρα θα μπορούσα να σας μιλήσω προσωπικά και να σας προτείνω το εξής. Μια κράτηση εκτός φυλακής είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Χρειάζεται ιδιαίτερο συντονισμό, χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών και σε σοφρονιστικά ζητήματα. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ε, συγκεκριμένες παραβιάσεις, να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή πόσο σοβαρά είναι τα εγκλήματα για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Γιατί όπως είπαμε η εγκληματικότητα δεν γνωρίζει σύνορα. Και έτσι κι αλλιώς την εγκληματικότητα δεν μπορούμε να την κλείσουμε ολόκληρη μέσα στις φυλακές. Η κυρία Ματιέ ρώτησε πώς οι υπάλληλοι, οι δεσμοφύλακες, όσοι εργάζονται στο σοφρονιστικό σύστημα, διατηρούν την ακαιρεότητά τους, παρά τις προσπάθειες που γίνονται μερικές φορές για δωροδοκία, διαφθορά κτλ. Όντως, στην Ισπανία και εγώ είχα προτείνει να μπορούμε να παρακολουθούμε τα τηλέφωνα. Οι νέες τεχνολογίες είναι αλήθεια ότι επιτρέπουν στους εγκληματίες που βρίσκονται στη φυλακή να εξακολουθούν να έχουν ε, συνδέσεις με τον έξω κόσμο. Μπορούμε όμως εμείς να σβήσουμε κάθε να αποκλείσουμε κάθε προσπάθεια ύποπτης επικοινωνίας. Δεν έχουμε πάντως πολλές περιπτώσεις. Μόνο σε μία φυλακή είχαμε πρόβλημα με τους ε, τρομοκράτες και ανακαστήκαμε και βάλαμε μια μονάδα η οποία ε, παρατηρεί και ελέγχει την τρομοκρατία από κοντά στις φυλακές. Τώρα, γιατί υπάρχουν λιγότερες γυναίκες από άντρες, πρέπει να σας πω σαν πρώτη σκέψη ότι οι γυναίκες συμμετέχουν πολύ λιγότερο σε εγκληματικές οργανώσεις από ότι άντρες. Και πιο συγκεκριμένα στη χώρα μου, το οργανωμένο έγκλημα που έχει να κάνει με την τρομοκρατία, με την τζιχάντ, οι φανατικοί έτσι κι αλλιώς δεν χρησιμοποιούν ε, τη γυναίκα για τέτοιου είδους δραστηριότητες εγκληματικές. Η κυρία Γιάλα Σέντερ αναφέρθηκε στην Κώστα Ντελσόλ και λέει ότι εκεί πάνε διακοπές οι μαφιόζοι. Και εμείς όμως έχουμε μαφία η ισπανική που δραστηριοποιείται στη Γαλλική κυρίως με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Πολλοί από τα ηγετικά της στελέχη βρίσκονται στη φυλακή. Δεν έχουν ε, παρετηθεί. Προσπαθούν ε, να εξακολουθούν να έχουν σύνδεση με την εγκληματική του οργάνωση. Γι' αυτό και εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε συντονισμό και προγράμματα βάσει των οποίων προσπαθούμε να συμφιλώσουμε τις δραστηριότητές μας και να χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο που έχουμε στη διάθεσή μας. Για παράδειγμα ζητάμε τη συνεργασία των πολιτών που αποδείχθηκε πολύτιμη στη Γαλλικία και πρέπει να συγχαρούμε τα άτομα τα οποία επιδεικνύουν τέτοιο θάρρος και μας βοηθούν να συλλάβουμε τους λαθρεμπορούς ναρκωτικών. 25.000 υπαλλήλους και προσωπικό έχουμε στο σοφρονιστικό μας σύστημα. Η εμπειρία μας με την τρομοκρατία μας έχει οδηγήσει να έχουμε μια καλή αναλογία κρατουμένων και ε, σοφρονιστικών υπαλλήλων. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε μία μία σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά θέλω να σας πω για τα θύματα ότι η νομοθεσία από το 2003 στην Ισπανία συμπεριφέρεται με ιδιαίτερο τρόπο στα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή της τρομοκρατίας, γιατί ζητάμε από τις τρομοκρατικές οργανώσεις και ε, της τρομοκρατίας να ζητούν συγνώμη από τα θύματα. πριν ε, καταλήψουν τη φυλακή. Πιο συγκεκριμένα, Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτηση της Πρόεδρου Αλφάνο, η φυλακή Βαλτεμόρο δεν είναι μια από τις πιο έτσι, εύκολες φυλακές μας, για να το πω απλά. Οι περισσότεροι από τους έγκλειστους, τους Ιταλούς, ζητούν να γυρίσουν στην Ιταλία βάσει της σύμβασης του Στρασβούργου. Είναι ο πρώτος νόμος της δημοκρατίας που θέλησε να δώσει κάποιες εγγύσεις στους κρατήμενους γιατί καταλαβαίνετε ότι περνούσαμε από μία περίοδο διαφορετική. Βλέπετε το 1974 υπήρχε αυτός ο νόμος, δεν μπορούμε να παρετηθούμε από αυτόν εξαιτίας του ιστορικού παρελθόντος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, να απαντήσετε γραπτά σε αυτούς που δεν μπορέσατε να απαντήσετε προφορικά. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω γραπτά σε όλες τις ερωτήσεις. Πολύ ωραία. Ε, πέντε λεπτά στην επόμενη μιλήτρια. Στον επόμενο μιλητή, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ε, σε πέντε δευτερόλεπτα θα απαντήσω ότι όλες μου σχέσεις, απαντήσεις έχουν σχέση με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Αν είχα πέντε δευτερόλεπτα θα λέγα αυτό. Επειδή όμως έχω παραπάνω χρόνο να πω τα εξή. Ένα λεπτό θα δώσω για κάθε ομάδα ερωτήσεων. Κύριε Γιακολίνο, μιλήσατε για συνοστισμό στις φυλακές. Ε, κοιτάξτε, θα παραμείνω λιγάκι γενικός εδώ. Πρόκειται για την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια. Δηλαδή, ε, η παραμονή στη φυλακή δεν είναι αυτή η τιμωρία. Η διάρκεια είναι η τιμωρία. Άρα δηλαδή αν δεν υπάρχει ε, για λόγους ασφαλείας να υπάρχει αυστηρή ποινή κάτω από το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να προστίθεται και η μεταχείριση στη διάρκεια. Και βεβαίως ο συνοστισμός στις φυλακές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω θα επανέλθω στο θέμα και στις άλλες ερωτήσεις που θα δώσω. Τώρα, απαντώ από κοινού ε, στην κυρία Μπορσελίνο και ε, στην κυρία Αλφάνο. Κοιτάξτε, εγώ επειδή έρχομαι από το βορρά της Ευρώπης δεν είμαι αρμόδιος προφανώς να μιλήσω για την Ιταλική νομοθεσία και το άρθρο ε, το 41 α που αναφέρατε, δεν ξέρω αν μπορώ να τοποθετηθώ επ' αυτού. Θέλω όμως να πω το εξής, ε, ότι τα νομικά και δικαστικά συστήματα δεν θα πρέπει να προκαλούν εχθρότητα. Δηλαδή όχι να σκληραίνουν τους ε, φυλακισμένους φυλακές. Ε, πρέπει η απόφαση να εκφράζει και την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Η ασφάλεια είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να εξισορροπείται με μια ανθρώπινη προσέγγιση για να αποδεικνύουμε ότι το κράτος είναι πάνω, πέρα και πάνω από ε, την βίαιη συμπεριφορά που επιδεικνύει άλλη πλευρά, οι εγκληματίες δηλαδή. Θέλω να επαναλάβω ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι δεν είναι και βέβαια φυλακές ε, ιδρύματα πολυτελούς διαβίωσης, ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά ούτε και να προκαλούμε ε, σκλήρινση των συναισθημάτων των ε, εγκλήστων. Προς τον κύριο Νιούτον Ντάν, θα ευχαριστώ πολύ που διευκρινίσατε το θέμα. Κοιτάξτε, εγώ ε, αν ήμουν στην Αστυνομική Ακαδημία ε, θα μπορούσα να μιλήσω πιο ελεύθερα. Εσείς αναφερθήκατε προηγουμένως στην άλμα Mater των πανεπιστημίων. Εγώ να σας μιλήσω προς τώρα για την δική μου την Ακαδημία. Ε, τώρα, αξιοπιστία και δίκαιο σύστημα, αυτά είναι σημαντικά, αλλά αν θέλετε να αναφέρω και ένα απλό παράδειγμα, το να αντιμετωπίσει κανείς το έγκλημα ε, σημαίνει ότι ε, προσπαθεί να το εξαλείψει. Νομίζω ότι το να μιλήσω για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό ε, θα ξεπερνούσε τις αρμοδιότητές μας. Εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Άρα δηλαδή όταν θέλουμε ε, να διαδώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει πρώτα να κοιτάμε τα του οίκου μας. Ε, αυτό έχει σχέση και με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έκανα μία μελέτη στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία ε, και μπορείτε να φανταστείτε γιατί διαλέξαμε αυτές τις τρεις φόρες διότι εκεί αναπτύσσονται τρομοκρατικές δραστηριότητες και πήραμε συνέντευξη κυρίως από παιδιά του σχολείου για να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι απόψεις τους για τη βία και προέκυψε σαφής διασύνδεση ανάμεσα στον κοινωνικό αποκλεισμό σε απλό επίπεδο με την τάση προς την βία. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την αρχική φάση αν θέλετε η διασύνδεση δεν είναι ανάμεσα σε μετανάστες και βία αλλά ανάμεσα στους κοινωνικά αποκλεισμένους και τη βία. Και μπορεί βέβαια κανείς να ε, πάει και σε άλλα επίπεδα, ε, σε ε, ήδη εγκλήστους ή σε ε, δυνάμει εγκλήστους σε αυτή την έρευνα πάντα. Εξάλλου πρέπει να αναθεωρούμε ε, και τα δικά μας τα συστήματα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το δικό μας εθνικό σύστημα είναι τέλειο και το ποινικό σύστημα είναι κάτι που δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε ακόμα και αν μας πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, εγώ Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αυτοκριτικοί, ε, να αναθερούμε λιγάκι τα συστήματά μας. Μιλήσατε και για την παγίδευση και εκεί ε, πρέπει να υπάρχει ισορροπία με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί κανείς να προσφέρει όλα τα δικαιώματα, αλλά να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο καλό του στόχου αφενός και στην προστασία των δεδομένων αφετέρου. Ξέρω ότι η παγίδευση τηλεφώνων χρησιμοποιείται ως μέσο σε ορισμένα κράτη-μέλη και ξέρω ότι δημιουργεί κάποια προβλήματα. Άλλα δύο θέματα να θίξω, γιατί ήδη μακρηγόρησα. Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό δώστε μου ακόμα να πω μόνο ε, προς ε, τον φίλο μου Ούλε όσον αφορά το PNR και το SWIFT ε, πέρα από αυτά που έχουμε ήδη πει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ούτε και εδώ, αλλά ε, το θέμα δεν είναι μόνο η αναλογικότητα, αλλά και η αποτελεσματικότητα. Είναι δηλαδή το PNR κάτι αποτελεσματικό ή μήπως επηρεάζει μόνο εκείνους που ελπίζει κανείς να συλλάβει με το PNR. Αυτοί όμως το ξέρουν το σύστημα και ξέρουν πώς να το αποφύγουν, παίρνουν άλλη διαδρομή. Τώρα, αναλογικότητα. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Στη γνωμοδότησή μας για τους ελέγχους ασφαλείας είπαμε και άλλοι ότι αυτοί οι έλεγχοι δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ε, πρέπει κανείς ε, να βλέπει όλα τα χαρακτηριστικά του σώματος ε, του ανθρώπου αρκεί να έχει ένα στίκ για να τα ελέγχει. Προς την Ισπανίδα βουλευτή να πω ότι εμείς έχουμε κάποια εμπειρία, έχουμε επισκεφτεί αρκετές φυλακές του κόσμου. Εγώ δεν το έκανα με την επαγγελματική μου ιδιότητα, πάντως θέλω να πω ότι και εδώ είναι απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία. Τα θύματα για να νιώθουν εμπιστοσύνη πρέπει να είναι ενημερωμένα, να εμπλέκονται να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους, δηλαδή ε, να μην δοθεί βέβαια από την άλλη η ε, ποινή, να μην σε αποδοθεί ποινή μετά από 10 χρόνια. Να τους αποδίδεται σημασία σε πάρα πολλούς τομείς, στις φυλακές, ε, στους υπόπτους, ε, στους εγκληματίες. Ξεκινώντας όμως με τους κρατικούς προπολογισμούς, πρέπει να πω ότι αυτή δεν είναι σε άμεση αναλογία με τα θύματα και σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ στο ότι πρόσφατα αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία εσείς στην οδηγία που εκπονήθηκε για τα θύματα. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε εδώ. Αν το θεωρείτε απαραίτητο, ε, θα ήθελα κατά τους επόμενους μήνες να σας να σας ε, συνοδεύσω σε ορισμένα σοφρονιστικά ε, καταστήματα στην Ιταλία για να δείτε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, περιμένουμε βέβαια τις γραπτές απαντήσεις του κυρίου που δεν είχε το χρόνο να απαντήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα θέματα που θέλετε να ρωτήσετε, αν, υπάρχουν, αν υπάρχει κάτι άλλο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι στις 17 ε, Σεπτεμβρίου ε, από τις 3 μέχρι 6.30 και στις 18 την επόμενη μέρα ολόκληρη τη μέρα. Σας υπενθυμίζω ότι η ΚΡΙΜ θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα με μια αντιπροσωπεία στη Σερβία. Θα έλεγα να φύγετε το στεμό των δυνατών ε, γιατί θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.